Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να συνεχίσουμε μετά τη διακοπή τη μεσημεριανή. Et je vous propose euh, d'en venir, euh, comme convenu, au point 19 de notre. Σας προτείνω λοιπόν να ασχοληθούμε με το σημείο 19 τη ημερήσια διάταξη. και να ακούσουμε την παρουσίαση του προγράμματο Εργασία 2010 τεσσάρων οργανισμών. Τεσσάρων οργανισμών, το οποίο το έργο έχει άμεση συνάφεια με την Επιτροπή μας. Πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας και το ε, Παγές Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θα ήθελα να πω σε εκπροσώπους των τεσσάρων οργανισμών ότι χθες κατά την ανταλλαγή, την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία της απαλλαγής προϋπολογισμού 2009 Η, εισηγήτριά μας από το ΕΛΚ αναφέρθηκε στις, στους τέσσερις οργανισμούς, όχι ειδικά, αλλά γενικά. Στα πλαίσια των παρατηρήσεων του ελεκτικού συνεδρίου που αφορούσαν οριζόντια όλους τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί διανύουμε μια φάση που το μοντέλο αυτό θα πρέπει να το αναπτύξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα που συζητάτε η ίδρυση τριών νέων οργανισμών, που δεν θα λέγονται οργανισμοί αλλά αρχές, αλλά θα έχουν παρόμοιες αρμοδιότητες ή καταστατικό και σχέση με την Επιτροπή, τα θεσμικά όργανα. Και κάνω μία των χθεσινών μας εργασιών και σχολείων για να σας ε, υπενθυμίσω ότι στις παρατηρήσεις σας, στις παρουσιάσεις που θα κάνετε εκπρόσωποι των τεσσάρων οργανισμών, θα μπορούσατε να σχολιάσετε και τις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Ακόμη και αν δεν είναι το μοναδικό θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης, ο σχολιασμός του ελεκτικού συνεδρίου μας ενδιαφέρει. Αν και επαναλαμβάνω, το κυρίως θέμα σήμερα είναι το πρόγραμμα εργασιών για το 2010. Θα ακούσουμε τη γενική παρουσίαση και μετά θα γίνει συζήτηση με τους παρόντες ευρωβουλευτές. Ναι. Θα ήθελα να είμαστε πειθαρχημένοι και να ακολουθήσουμε τη σειρά που προβλέπει η μερίσια διάταξη. Οπότε πρώτα θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Θα ακούσουμε τον κύριο Γιού Κατάκαλα, Χρόνου φίδου, παρακαλώ. Αλλά φαντάζομαι το ξέρετε, αυτό δεν χρειάζεται να μακρηγορήσετε. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ πάλι. Έχετε το εγγραφό μου, δεν θα το διαβάσω. Ούτε θα παρουσιάσω μία παρουσίαση με διαφάνειες, με PowerPoint, η οποία είναι ακριβώς ίδια με αυτά τα οποία περιέχει το έγγραφό μου. Θα τονίσω όμως τα σημεία κλειδιά του προγράμματός μας 2009-2010. Ασφαλώς ε, βεβαίω, ορισμένα στοιχεία έχουν σηματωθεί στο πρόγραμμα του 2010 από το 2009. Όπως όλοι ξέρετε, ε, οι συνθήκες εργασίας, η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί με νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα. Βεβαίως ε, το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο είναι σημαντικό, αλλά δεν επαρκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο φέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη σωστή εφαρμογή επίσης η Κομισιόν αλλά και τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλες αρμοδιότητες. Πρέπει εμείς να προωθήσουμε αυτό το πλαίσιο και σήμερα το πρωί μιλήσαμε για το ρόλο της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας και χάρηκα που άκουσα από την Πρόεδρο ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί τώρα σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας να πιστοποιήσει να εγκρίνει δηλαδή ε, τις συμβάσεις ε, τους, ε, της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας. Ε, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, το ILO, έχει εκδώσει πάρα πολλές σύγχρονες και επίκαιρες συμβάσεις για το χώρο εργασίας. Έχω στο παρελθόν εργαστεί 25 χρόνια για την οργάνωση αυτή και αυτή την εμπειρογνωμοσύνη φέρνω εγώ στην Επιτροπή σας. Από αυτό το, το υπόβαθρο δηλαδή ομιλώ. Ε, έχουμε έναν ιδιαίτερο καθήκον στο Ίδρυμα του Μπιλμπάου, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό που είναι στο Μπιλμπάου, ε, να οργανώσουμε εκστρατείες για την ασφάλεια και την υγεία. Ξέρετε, είσαστε ενήμεροι για τις τρεις αυτές εκστρατείες μας ε, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, έχουν δηλαδή προτεραιότητα ε, για όλες τις δραστηριότητε που αφορούν την εφαρμογή των ε, συστάσεων και των οδηγιών. Η τελευταία μας εκστρατεία συμπεριέλαβε ένα συνέδριο με 500 συμμετέχοντες με υπουργούς ε, από τη Σουηδική Προεδρία και συζητήσαμε το θέμα της αξιολόγησης κινδύνων και είχαμε λόγω αυτής της εκστρατείας μια πάρα πολύ καλή ε, δημόσια παρουσίαση και ε, δόθηκε πολύ θετική δημοσιότητα σε εργασίες του οργανισμού μας. Τονίσαμε επίσης σε αυτό το συνέδριο ότι κάθε μέρα, κάθε μέρα ε, 167.000 άνθρωποι ε, χάνονται, σκοτώνονται δηλαδή, ε, λόγω της ανασφάλειας ε, στην εργασία, λόγω προβλημάτων και ατυχημάτων στην εργασία. Σε, ε, σε ένα αεροπλάνο, αν πέσει ο Θεός να φυλάει ένα αεροπλάνο, σκοτώνονται ας πούμε 200 άνθρωποι. Εμείς όμως ε, μέσα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό τον τεράστιο αριθμό των θανάτων, 167.000. Είναι λοιπόν πιεστική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε αυτό τον αριθμό. 450 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μέρα ε, στην εργασία. Ο Σουηδός Υπουργός λοιπόν μα είπε ότι ένας από τους τρεις ανθρώπους ε, ε, είναι άνεργος. Ένας από τους τρεις, ένας στους τρεις, 30% και κάτι. Ε, η... Στην Ισπανία είναι 20% η ανεργία, περίπου, λίγο πολύ. Αλλά ένας στους τρεις στη Σουηδία, καταλαβαίνετε πόσο μπορεί αυτό το ποσοστό να επηρεαστεί από τις συνθήκες στην εργασία, από το management της εταιρεία και τους ε, συναφείς παράγοντες. Αυτά, με αυτά λοιπόν ασχολούμεθα σε όλους τους τομείς της ε, οικονομίας, διατομεακά. Το δεύτερο θέμα κλειδί που θέλω να τονίσω είναι μια κληρονομιά από το όλο θέμα της αξιολόγησης κινδύνου. Μπορεί να έχετε ακούσει για την Επιτροπή Στόιμπερ, η οποία προτείνει την μείωση του διοικητικού κόστους, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι εμείς έχουμε μια λύση στα χέρια μας. Καταρχάς, η υποχρέωση η υποχρέωση ε, μιας μελέτης αξιολόγησης κινδύνου μπορεί να διευκολυνθεί για μια μικρομεσαία επιχείρηση και να γίνει online, δηλαδή μέσω του διαδικτύου ή και τηλεφωνικά. Αντί λοιπόν να πληρώσει έναν εξωτερικό σύμβουλο 10.000 ευρώ για να του υποβάλει μια μελέτη εξολόγηση κινδύνου, μπορεί ο μικρομεσαίο επιχειρηματία να χρησιμοποιήσει ή το διαδίκτυο ή το τηλέφωνο. Ορισμένοι πιστεύουν το θέμα αυτό είναι δύσκολο, αλλά εμεί πιστεύουμε ότι είναι εφικτό ή, είτε εφαρμόζοντάς του στην αρχή σε ένα πολύ μικρό περιορισμένο επίπεδο και μπορεί να χρειαστούμε με επιπλέον πόρους, ε, όχι πολύ σημαντικούς δηλαδή, για αυτή την εφαρμογή. Και δεύτερον, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τον τριμερή μηχανισμό δηλαδή ε, εργοδότες, εργαζόμενοι και δημόσιο, κυβέρνηση δηλαδή, να διατεθεί ε, ένα, μια πίστοση για ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην Ολλανδία. 150.000 ε, έχουμε εμείς βεβαίως ε, ε, ευρώ προϋπολογισμό για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η Ολλανδία που εφαρμόζει ένα πιλωτικό πρόγραμμα έχει ήδη διαθέσει 5 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Όμως, Όσον αφορά τη μελέτη για το, ε, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους αναδυόμενους κινδύνους, θα έχουμε τα αποτελέσματα σε μια έκθεση την Άνοιξη που θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αναδυόμενους κινδύνους. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι κίνδυνοι. Καταρχάς, όσον αφορά τις, ε, τα, ειδικές, άτομα με ειδικές ανάγκες ε, και, και αναπηρίες ποιοι είναι οι λόγοι, ποιε είναι οι αιτίες. Ε, οι αιτίες. Στη Φιλανδία έχουμε ποσοστά 46% ε, σε γυναίκες δηλαδή που είναι αποδέκτες ε, επιδομάτων αναπηρίας και γενικά βοηθημάτων επειδή είναι άτομα με ειδικέ ανάγκες. Είναι λοιπόν ε, και συνήθως γυναίκες που έχουν συνταξιοδοτηθεί, αλλά είναι πολύ ψηλό το ποσοστό αυτών που λαμβάνουν αυτά τα επιδόματα αναπηρίας. Και τέλος, δια, δια, όσον αφορά τη στρατηγική του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω ότι πρέπει να τονίσει μόνο την απασχόληση. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι όμως οποιαδήποτε απασχόληση. Μία απασχόληση που θέλουμε να είναι ποιοτική, αναβαθμισμένη, να δίνει τη δυνατότητα διαβίου εκπαίδευσης και, και συνεχούς απασχόλησης, εργασίες δηλαδή, μια ποιοτικά αναβαθμισμένη εργασία. Αν το επιτύχουμε αυτό, τότε θα επιτύχουμε να προωθήσουμε ένα, ένα την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πλήρη παρουσίαση που μας κάνατε. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Βουλγαρέλη από το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και θα συνεχίσουμε μετά. Κυρία Βουλγαρέλη, παρακαλώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θέλω να πω ότι με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Επιτροπή σας για να σας ενημερώσω για τα επιτεύγματα και τις δραστηριότητες του ΣΕΝΤΕΦΟ το 2009 και τι προβλέπουμε να κάνουμε το 2010. Καταρχάς θέλω να κάνω μία δήληση. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μεμονωμένων ατόμων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη σημερινή κρίση και να ανταποκριθούν στις αυριανές εργασίες είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οι δεξιότητες, η μόρφωση και η εκπαίδευση βρίσκονται στην καρδιά της ε, στρατηγικής της Λισαβόνας, της στρατηγικής απασχόλησης βεβαίως. Και βεβαίως επίσης βρίσκονται στην καρδιά της έκθεσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στρατηγική του 2020. Η οικονομική κρίση σήμερα έχει τονίσει πόσο χρειάζονται οι δεξιότητες στην Ευρώπη. Μία μελέτη την οποία έκανε το ΣΕΝΤΕΦΟΠ σε συνεργασία με την Σουηδική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 συνεπέρανε ότι θα πρέπει να, προβάλλ, να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για να διατηρήσουμε το εργατικό μας δυναμικό, ένα σημαντικό κεφάλαιο και για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις, εργασί... τις εργασίες τους, το κεφάλαιο της εργασίας τους. Για να γίνει αυτό πρέπει να αναζωογονηθεί η οικονομία και ε, να χρησιμοποιηθούν ε, ε, ευέλικτες μορφές εργασίας, παραδείγματο χάρη με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου, μερική επασχόληση κλπ. Είμαστε ένα νέο κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης. Γι' αυτό μία από τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές μας είναι να παρουσιάζουμε προβλέψεις για τις, τις ευρωπαϊκές ανάγκες σε δεξιότητες και στην κατάρτιση. Το ΣΕΝΤΕΦΟΠ τα τελευταία χρόνια είναι η βασική πηγή παροχής πληροφοριών για τις ανάγκες αυτές ε, της εργασίας, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Εκπαίδευσης σε νέες εργασίες, σε νέες μορφές εργασίες και αυτή η ανάγκη συνεχούς ε, ενημέρωσης ε, περιέχεται και στο έγγραφο της Κομισιόν. Το Φεβρουάριο του 2010 θα παρουσιάσουμε τις καινούργιες προβλέψεις μας που έχουν λάβει υπόψη την οικονομική κρίση. Έχουμε βεβαίω συνεργαστεί με η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και θα διοργανώσουμε ε, ένα συνέδριο όπου θα σας καλέσουμε βεβαίω και θα χαρούμε να σας δούμε. Επίσης έχουμε συνεργαστεί και με τον εισηγητή κύριο Όλε Κρίστενσεν, ο οποίος ανέλευε την πρωτοβουλία να διοργανώσει μια κοινή συνεδρίαση μεταξύ ΣΕΝΤΕΦΟΠ και της Επιτροπής σας και αυτή η συνεδρίαση θα γίνει στις 2 Μαρτίου. Επιτροπή Απασχόλησης και ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Θα είναι λοιπόν μια θαυμάσια ευκαιρία να συζητήσουμε τις προβλέψεις μας και τις προτάσεις μας και να ακούσουμε τις απόψεις σας. Λοιπόν, θα σας δώσω τώρα ορισμένες ε, προβλέψεις για το 2020. 80 εκατομμύρια νέες ευκαιρίες εργασίας πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν μέχρι το 2020. Πρέπει όμως να προσέξουμε τις εργασιακές τάσεις. Τι είδους εργασίες. Οι εργασίες αυτές απαιτούν καινούριε, αναβασμισμένες δεξιότητες και υψηλότερα προσόντα. Αυτά θα τα συζητήσουμε βεβαίως στην κοινή συνεδρίαση που θα κάνουμε. Οι απαιτήσει σε δεξιότητες στο μέλλον δείχνουν ότι θα πρέπει η Ευρώπη να επενδύσει σημαντικά στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη όχι μόνο για τη νέα γενιά αλλά και για τους όριμους εργαζόμενους, τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους. Πολλά πράγματα συμβαίνουν που καθιστούν την εργασία πιο ευέλικτη αλλά και την πρόσβαση στην αγορά για να μπορέσουν να βοηθήσουν ε, εκατομμύρια πολίτες μας. Ενθαρρύνουμε την κινητικότητα και την εκπαίδευση των εργαζομένων και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχει συνεργαστεί πάρα πολύ στενά με τους αρμόδιους φορείς. Η δεύτερη μεσοπρόθεσμη προτεραιότητά μας είναι να παρουσιάσουμε τα απαραίτητα στοιχεία πάνω στα οποία θα στηριχθεί η ευρωπαϊκή πολιτική ανάπτυξης και επαγγελματικής ε, κατάρτισης. Ε, σύμφωνα ε, με αυτά που ζήτησε το Συμβούλιο από εμά, το ΣΕΔΕΦΟΠ παρακολουθεί και υποβάλλει μία έκθεση κάθε δύο χρόνια για τα κράτη-μέλη, μία έκθεση δηλαδή για το πώς έχουν υλοποιήσει τις προτεραιότητες αυτές. Και στην Μπρούζ το Δεκέμβριο το 2010 θα παρουσιάσουμε μια συνολική έκθεση αξιολόγησης της διαδικασίας της Κοπενχάγης, που αφορά βεβαίως τη διαβίω ανάπτυξη, ε, τη διαβίω εκπαίδευση. Η προηγούμενη μας ολοκληρωμένη έκθεση είχε τον τίτλο ε, «Συνεχής παγίωση σε, μια, σε ένα κλίμα αλλαγής» και κάλυπτε την περίοδο 2008-2010. Αυτή ήταν η προηγούμενη έκθεση. Η επόμενη θα παρουσιαστεί το Δεκέμβριο. Θα ήθελα επίσης να, να σας ενημερώσω για την, ε, τις νέες εξελίξεις στην μεταρρύθμιση των, ε, Ευρω... της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. Η, όσον αφορά τα προσόντα. Το νέο πλαίσιο ευρωπαϊκών προσόντων έχει βασιστεί στις προτάσεις του ΣΕΝΤΕΦΟΠ και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ έχει δημιουργήσει καινούργια εργαλεία, καινούργια μέσα εφαρμογής, υλοποίησης του προγράμματος αυτού. Το 2009 ακολουθήσαμε τις συστάσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Επαγγελματική κατάταση ΕΚΒΕΤ ε, και συστήσαμε και ένα ε, πλαίσιο αναφοράς ε, Εκπονήσαμε λοιπόν τα απαραίτητα και δημιουργήσαμε τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουμε και να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε τα ευρωπαϊκά προσόντα έτσι ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μελέτης και αξιολόγησης των ευρωπαϊκών ε, επαγγελματικών προσόντων. Έχουμε επίσης ε, αναπτύξει ε, δημιουργήσει ένα φάκελο για τις δραστηριότητες μας από το 2005 σε πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες και 25 εκατομμύρια ε, χρήστες του διαδικτύου έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας, ε, έχουν απαντήσει σε ερωτηματολόγια και χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες μας. Αυτή τη στιγμή πλέον υπάρχει ένα πρότυπο ευρωπαϊκό που CV, ε, ευρωπαϊκής, ε, ευρωπαϊκού βιογραφικού. Το ευρωπαϊκό βιογραφικό λοιπόν είναι άλλη μια επιτυχία που εξελίχθηκε με τη βοήθεια του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Τα μέσα, τα εργαλεία τα οποία προσπαθούμε εμείς να δημιουργήσουμε στοχεύουν στην αύξηση της κινητικότητας ε, των, και της ευελιξίας των Ευρωπαίων εργαζομένων Είχατε, σας είχαμε αποστείλει ένα συνοπτικό σημείωμα για τις δραστηριότητες μας ε, του 2010. Δεν θα τα επαναλάβω όλα αυτά, απλώς θα τονίσω ότι θα προσέξουμε ιδιαίτερα τις δεξιότητες, ε, την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ανάπτυξης Προσόντων, και θα, θα παρακολουθήσουμε επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στην ανάπτυξη των ιατρικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Έχουμε βεβαίως το διοικητικό μας συμβούλιο όπου εκπροσωπείται η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και συνεργαζόμαστε με, τις, με τα αδελφά ιδρύματα. Έχουμε συμφωνίες, συνεργασίες με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ε, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Ε, με το οποίο συνεργαζόμαστε σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και ε, εργασιακών σχέσεων. Α, και επίσης τώρα θα αρχίσουμε μια νέα συνεργασία, μια συνεργασία με το νέο Ίδρυμα για την ε, ισότητα του φύλων. Όλες μας οι δραστηριότητες βασίζονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να σας παραθέσω ένα απόσπασμα από μια έκθεση αξιολόγησης που έγινε για μας, για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ ε, και που κατόπιν εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει λοιπόν το σχέδιο έκθεσης αυτό αξιολόγηση, ότι το ΣΕΝΤΕΦΟ προσφέρει φέρει μεγάλη αξία, ε, έχει μια προσφορά μέγιστης αξίας δηλαδή στο, στις αρμοδιότητες με τις οποίες ασχολείται και ε, αυτή λοιπόν το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης μας έκανε λίγαν υπερήφανους για την εργασία που κάνουμε. το ΣΕΝΤΕΦΟΠ χρησιμοποιεί ε, ένα, τον προϋπολογισμό του για να καθορίσει τις εφικτές ε, δραστηριότητες. Ε, αυτά δηλαδή τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και πιστεύω ότι έχουμε πράγματι εφαρμόσει ε, τις ε, προτάσεις του, του, ελεγκτικού συνεδρίου να χρησιμοποιούμε ξύπνιους, έξυπνους όπως λέμε, δείκτες όσον αφορά τη σωστή εφαρμογή του προϋπολογισμού και των λογιστικών και θέλουμε στο μέλλον όχι μόνο να μπορούμε να μετρήσουμε σαφώς την παραγωγή μας, αλλά και την επίπτωση την οποία έχουν οι δραστηριότητές μας. Έχω ένα μεγάλο κατάλογο δικτών, μετρήσιμων δικτών, τους οποίους χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε τον οργανισμό μας και όλα αυτά θα περιληφθούν στην ετήσια έκθεσή μας. Εν πάση περιπτώσει, κατα, καταλήγω ότι έχουμε μετρήσιμα εργαλεία για να ελέγχουμε την απόδοσή μας και την παραγωγή μας. Επίσης, σεβόμαστε τις διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις μεταφορές, τα carry-overs από το 2008 στα επόμενα χρόνια. Δεν έχει το ελεγκτικό συνείδριο τίποτα να παρατηρήσει από αυτού. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε και τα ελέγχουμε εις βάθος. Και πάλι λοιπόν σας παραθέτω ένα απόσπασμα από την εξωτερική αξιολόγηση όπου ο αξιολογητής λέει ότι το βασικό σημείο κλειδί για την μέγιστη αποτελεσματικότητα κόστους έγκυται στη σωστή εποπτεία και στο σωστό έλεγχο του ετησίου προγράμματος. Το ετήσιο πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα και σωστή εφαρμογή του καλύπτει και το θέμα του ελέγχου των δραστηριοτήτων, ε, ιδίω όσον αφορά την εξέβρεση λύσεων σε προβληματικά θέματα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την υπομονή σας και το χρόνο σας και θα ήθελα να καλέσω την κυρία Πρόεδρο να μας επισκεφθεί και προσβλέπω με μεγάλη χαρά στην ε, ε, κοινή μας συνεδρίαση ε, στις 2 Μαρτίου που θα κάνουμε με την Επιτροπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε και ευχαριστούμε και για την πρόταση συνεργασία για τους επόμενους μήνες. Τρίτη παρέμβαση. Εξ του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας. Τον Ο κύριος Γιώρμα Καρπίνεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπέρες. Είναι μεγάλη η χαρά μου ως εκπροσώπου του Eurofound να βρίσκομαι εδώ για μια ακόμα φορά. Έχουμε ήδη μοιράσει γραπτό ε, υλικό το οποίο αναφέρεται σε μια εκτεταμένη περίληψη των δραστηριοτήτων μας και βεβαίως οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να έχετε το πλήρες πρόγραμμά μας για το 2010. Ε, έχουμε όλη την τεκμηρίωση την οποία χρειάζεστε. Ε, όμως τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια έτσι ώστε να ε, δώσω μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση. Ε, πρέπει να πούμε ότι η Eurofound την προηγούμενη χρονιά είχε την, ε, τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο όλες οι αναφορές στις έρευνές μας και στα προγράμματά μας ήταν εξαιρετικά θετικές από όλα τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Επίσης, εκλήθημε να συμμετάσχουμε σε πολλές ομάδες εργασίας και προσβλέπουμε και σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν 20 ομάδες εργασίας ε, σχετικά ε, με την δημιουργία θέσεων εργασίας, σχετικά με την βελτίωση των θέσεων των συνθηκών εργασίας, ε, και διάφορα άλλα ε, θέματα και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους ε, δείκτες όσον αφορά την, τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης που θα περιλαμβάνουν δηλαδή επιπλέον δείκτες όσον αφορά την επεγγελματική ολοκλήρωση κλπ. Το 2010 είναι το δεύτερο έτος του παρόντος μας προγράμματος και ελπίζουμε ότι θα μας δώσει την ε, δυνατότητα να ολοκληρώσουμε αυτά που ξεκινήσαμε το 2009. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε τρεις ε, ε, μελέτες η πρώτη ήταν ε, η European Company Survey, ε, η δεύτερη, δηλαδή για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η δεύτερη ήταν ε, για την ευελιξία στην Ευρώπη και η τρίτη ήταν μια μελέτη επιτόπου, η οποία ξεκίνησε στην αρχή του 2009, δηλαδή πάνω ακριβώς στο αποκορύφωμα της κρίσης, που ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα ευρήματα εκεί ήταν αρκετά σημαντικά. Δηλαδή, στην ουσία μας έδειξαν τα ευρήματα ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καταφέρνουν να προσαρμοστούν ε, στο νέο περιβάλλον. Ο διάλογος, ο κοινωνικός διάλογος ε, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φαίνεται ότι είναι, εξακολουθεί να είναι καλά στην υγεία του και αυτός ε, ο μηχανισμός είναι κάτι πολύ θετικό. Ε, επίσης είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, μελέτη ε, σχετικά με την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη και μια ειδική έκθεση σχετικά με σύγκριση της αντίληψης ε, ποιότητας ζωής ε, το Σεπτέμβριο του 2008 ε, σε σχέση με την περίοδο μετά την κρίση. Ποιότητα ζωής λοιπόν και αντίληψη της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων και εκεί τα ευρήματα ήταν πολύ σημαντικά. Φάνηκε σαφώς ότι υπήρξε αντίκτυπος της κρίσης στην ε, ε, ζωή των ε, Ευρωπαίων και επίσης ταυτοχρόνως διαπιστώσαμε μείωση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων στα πολιτικά συστήματα, στα οικονομικά συστήματα κτλ. Επίσης, στο 2009 προετοιμαστήκαμε για την πέμπτη ετήσια έρευνα όσον αφορά τις συνθήκες ε, εργασίας. Δημιουργήσαμε τρία παρατηρητήρια, δημοσιεύσαμε ε, ε, πάρα πολλά άρθρα, συγκριτικές μελέτες, συγκριτικά στοιχεία και γενικώ απέρευσαν από τα παρατηρητήρια 10 συγκριτικέ μελέτες σχετικά με την αυτοεπιχειρηματικότητα, σχετικά με του ελεύθερου επαγγελματίες κλπ. Ε, και, ε, φέτος στο ε, έχουμε ένα παρατηρητήριο σχετικά με την αναδιάρθρωση της ε, οικονομίας και κυρίως όσον αφορά αναδιαρθρώσεις ε, σε βιομηχανίες. Ακριβώς αυτό το θέμα αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά σημεία μελέτης μας για το 2009. Συνεργαζόμαστε επίσης όλο και περισσότερο και με καλύτερο τρόπο, πιο εμβαθυμένο, με πολλές άλλες ε, ε, οργανώσεις, με τις υπηρεσίες της Κομισιόν, με τη Eurostat φυσικά ε, και, και με άλλους οργανισμούς, με την κυρία Βουλγαρέλη ας πούμε έχουμε στενά συνεργαστεί. Τώρα κάποια μεμονωμένα παραδείγματα αποτελέσματος. Πέρσι, ε, όσον αφορά την ε, παρακολούθηση αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων και κυρίως βιομηχανιών, ε, εμείς εκπονήσαμε τριμηνιές, διμηνιές, τριμηνιές και τετραμηνιές εκθέσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις Επίσης ε, καταφέραμε να αντιδράσουμε πάρα πολύ γρήγορα με εκθέσεις όσον αφορά ε, ε, τομείς σε ύφεση. Τώρα για τη βιομηχανία γενικά κάναμε μελέτη σχετικά με την πορεία της βιομηχανίας σε σχέση με την συνολική πορεία της οικονομίας σε περιοχές της Ευρώπης. Επίσης ε, δημιουργήσαμε, ε, δημοσιεύσαμε ε, τον πρώτο ευρωπαϊκό κατάλογο των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών με τα αποτελεσματά τους. Τώρα τον Μάρτιο θα είμαστε σε θέση να δώσουμε τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης για τις επιχειρήσεις για να δούμε πώς ακριβώς αντέδρασαν οι επιχειρήσεις σε, αυτόν σε αυτήν την ε, ε, οικονομική κρίση. Επίσης κάνουμε μελέτες σχετικά με, τους, ε, με τα άτομα με αναπηρία, εργαζόμενους με ειδικά προβλήματα. Και όλα αυτά τα κάναμε ήδη μέσα στο 2009. έχουμε ένα ε, πλήρες πρόγραμμα εργασίας ε, και βάσει αυτού του προγράμματος ε, έχουμε προχωρήσει σε μελέτες. Προσπαθούμε μακροσκοπικά να δούμε την αγορά εργασίας της Ευρώπης ε, αγορά εργασία η οποία βεβαίως βρίσκεται σε πλήρη αναταραχή ε, αυτή την εποχή. Όσον αφορά την flex security, βεβαίως ε, είναι ευελιξία και ασφάλεια, βεβαίως είναι ένα από τα κεντρικά στοιχεία που μας απασχολούν έτσι ώστε να αξιολογήσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, ε, επίσης βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για τις συνθήκες εργασίας, ε, θέλουν να ασχοληθούν με θέματα όπως είναι η έλλειψη θέσεων απασχόλησης, όπως είναι η κινητικότητα κτλ. Τώρα στην εικόνα, στη διαφάνεια που βλέπετε στα δεξιά ε, προσπαθούμε να, έχουμε, ε, προσπαθούμε να κάνουμε μελέτες ε, όσον αφορά ας πούμε την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της αηφόρου κοινωνικής προστασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειες και την εργασία, για οικονομικούς, κοινωνικούς και για, για οικονομική πολιτιστική ε, και κοινωνική ένταξη των ε, ε, μεταναστών για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας κτλ. Όλα τα αποτελέσματα όλων αυτών, την, τον όλα αυτά τα αποτελέσματα των μελετών θα παρουσιαστούν σε, ειδικό σεμινάριο εδώ στις Βρυξέλλες το Σεπτέμβριο του 2010. και επίσης τώρα προετοιμαζόμαστε ε, για την δεύτερη μεγάλη μελέτη που θα γίνει του χρόνου του 2011 για την ευρωπαϊκή ποιότητα ζωής. Και επίσης θα έχουμε κι άλλα ε, κεντρικά αποτελέσματα όσον αφορά τις τάσεις ε, της απασχόλησης στην Ευρώπη Έχουμε δημιουργήσει το, το σύστημα European Jobs Monitor ε, για την παρακολούθηση των, ε, ε, της απασχόλησης και των, των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Εκεί βλέπουμε, παρακολουθούμε από κοντά τις απώλειες θέσεων εργασίας κλπ. Κάθε έξι μήνες ε, θα κάνουμε αναφορά ε, σχετικά με αυτό το EJM, το European Jobs Monitor. Όσον αφορά τώρα τη, τις ε, καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και την μεγαλύτερη παραγωγικότητα μέσω εταιρικών σχέσεων, εκεί βλέπουμε τομεακά τους κοινωνικούς ε, εταίρους ε, μέσω αντιπροσωπευτικών μελετών, μετά από αίτημα μάλιστα σχετικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε τις βιομηχανικές ε, σχέσεις και την αηφορία, την οικονομική κρίση και την εξέλιξη της εργασίας και της απασχόλησης όσον αφορά μη τυποποιημένες μορφές εργασίας, καθώς επίσης και τις διασυνδέσεις μεταξύ ποιότητας εργασίας και απόδοσης. Ναι, όσον αφορά τώρα τον τομέα της προώθησης της κοινωνικής ε, ε, ε, της ε, κοινωνικής ολοκλήρωσης και της αηφόρου και αποτελεσματικής κοινωνικής προστασίας. Εκεί εντάσσονται οι πρωτοβουλίες των εταιριών έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στην απασχόληση και την περίθεψη, η οικονομική κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών κλπ. Ε, όσον αφορά τώρα την, ε, τον προϋπολογισμό μας, ε, κατανοούμε ότι σε περιόδους κρίσεως τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα. Όπως είπα και προηγουμένως, βλέπουμε ότι βάσει λόγω μάλλον της αναταραχής στις αγορές διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος στρέφεται προς καλύτερα προνοιακά ε, συστήματα. Ε, ε, όσον αφορά τώρα τον δικό μας προϋπολογισμό για την Eurofound, το 2010 θα έχουμε 20.340.000 συμπεριλαμβανομένου και του IPA ε, όσον αφορά τώρα τις, ε, ε, τους ανθρώπινους πόρους, εμείς προσπαθούμε να έχουμε μια οργάνωση εργασίας βάσει μόνιμων συνεργατών. Ε, τώρα, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάποιες ε, μεταφορές ποσών, κάποια κάποια carry-overs, ε, τα οποία είναι λογικά εάν λάβει κανείς υπόψη τον, προϋπο, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και αυτές τις έρευνες, οι οποίες δεν ολοκληρώνονται πάντα τη στιγμή που πρέπει. επανέρχομαι στο θέμα των ε, των ανθρωπίνων πόρων. Εκεί εστιαζόμαστε ε, σε πολυτομιακά και εγκάρσια προγράμματα, ομάδες μάλλον για πολυτομιακά και εγκάρσια προγράμματα, ε, τα οποία στηρίζονται από οργανισμούς ευέλικτους. Όσον αφορά τώρα ε, την παρακολούθηση και τις αξιολογήσεις. Ε, έχουμε ένα πολιετές ε, πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης και υπάρχει και η ενδοοργανική αξιολόγηση. Έχουμε το ε, EPMS, Eurofound Performance Monitoring System, ε, το οποίο μετρά την πρόοδο της ε, Eurofound όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και που έχει λειτουργήσει σε τετραετή βάση. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και επομένως νομίζω ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα και βεβαίως ε, ε, εξεκολουθούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το ε, PMS. Τέλος, αλλά καθόλου Ελλάσσον, έχουμε βεβαίως εδώ και την παρουσία μας στις ε, Βρυξέλλες. Ε, κάθε τόσο ζητούμε από το γραφείο μας των Βρυξελών διάφορες εξυπηρετήσεις και διάφορες υπηρεσίες, τις οποίες με χαρά μας προσφέρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, και περνάμε στην τελευταία παρουσίαση από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συγγνώμη για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης και πριν δώσω το λόγο στην αρμόδια του Ιδρύματος αυτού, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι έχουμε στην αίθουσα τρεις ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, όπως διορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το κέντρο αυτό. Την κυρία Σάρα Πάρκινγκ, τον κύριο Παλοκρασά και τον κύριο Μεζιέρ. Μας τιμά η παρουσία τους σήμερα εδώ στη συνεδρίασή μας. Ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Μαντλέν Σερμπάν, για την τελευταία αυτή παρουσίαση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματική Κατάρτισης. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτά. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι είναι μεγάλο προνόμιο για μένα να βρίσκουμε εδώ στην πρώτη μου αυτή ακριβώς ε, δραστηριότητα αναφοράς και ενημέρωσης του Ιδρύματός μας στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το τι έχουμε κάνει και το 2009 και τους στόχους μας για το 2010 και να σας ε, δώσω μία ανοιχτή πρόσκληση, να προσφέρω μία ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σας να μας επισκεφθούν στο Τωρίνο για να ενημερωθούν επί τόπου το Ίδρυμά μας λειτουργεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το τονίσω για να σας εξηγήσω ότι από αυτήν την άποψη είμαστε μοναδικοί όσον αφορά τη σύγκριση με τα άλλα κέντρα και ιδρύματα. Δουλεύουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ Είμαι πολύ ευγνώμων στα ευρωπαϊκά ε, θεσμικά όργανα τα οποία αποφάσισαν ότι το, ο βασικός στόχος της ανάπτυξης είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Δηλαδή, να υποστηρίξουμε τις γειτονικές ε, και συνεργάτιδες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους μέσω της εκπαίδευσης, ε, της κατάρτισης ε, και των συναφών προγραμμάτων για να μπορέσουν οι χώρες αυτές αναπτύσσοντας την επαγγελματική κατάρτιση να ωφελήσουν τους πολίτες μας. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματική Κατάρτισης εκπονεί πολιτικές, όχι όμως ε, για να ε, δημιουργήσει νέες διαδικασίες, αλλά για να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών των γειτονικών χωρών. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου και του κοινωνικού κεφαλαίου είναι τα βασικά ε, ζητήματα, οι βασικοί τομείς που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη και να αναβαθμίσουν τις ε, χώρες αυτές και τις σχέσεις με τις χώρες αυτές στο πλαίσιο εξωτερικής συνεργασίας. Η βασική τομή τους οποίους τονίσαμε το 2009 ήταν η υποστήριξη προς την Κομισιόν των εξωτερικών πολιτικών της που αφορούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Για να το επιτύχουμε αυτό, συνεργαστήκαμε με τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ε, την Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων, τη ΡΕΛΕΞ, αλλά και με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Και ε, κατόπιν ετήματος με, της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης προετοιμάζουμε τις υποψήφιες προσένταξη χώρες ε, συμπεριλαμβανομένης ε, και της Τουρκίας ε, να, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και να βοηθήσουμε την, ε, το, ώστε το Ταμείο αυτό να έχει θετικές επιπτώσεις στις, χώρες, στις αποδέκτες χώρες. Πρέπει λοιπόν να αναφερθώ ε, και στο πρόβλημα της ε, μετανάστευσης We are not working... και της παράνομης μετανάστευσης. Ε, δεν θέλουμε να ενισχύσουμε ε, την ε, μετανάστευση χωρίς κανένα ιδιαίτερο σκοπό. Θέλουμε την να ενισχύσουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Γι' αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε την κινητικότητα του, του εργατικού δυναμικού ώστε να βοηθηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτός λοιπόν από την, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Στην περιοχή ε, Μέντα, την περιοχή δηλαδή της Ανατολικής Μεσογείου και συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Εκεί υποστηρίζουμε την ανάπτυξη επιχειρήσεων και σε αυτή την περιοχή του κόσμου η επαγγελματική κατάρτιση δεν την περιλαμβάνει μόνο και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ε, καλύπτει και την τριτο, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσω της ad hoc ε, συντονίζουμε την ενίσχυση της ενισχύσης και τη βοήθεια που προσφέρουμε για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων μέσα στα πλαίσια της περιεχόμενης βοήθειας. Η παρεχόμενη λοιπόν βοήθεια μέσα στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να εφαρμόζεται ε, μέσω των βέλτιστων προγραμμάτων. Ο βασικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε τον προγραμματισμό της εξωτερικής βοήθειας με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αφού πρώτα διαπιστώσουμε τι ανάγκες έχουν οι αποδέκτριες χώρες όλες οι 30 ε, χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, εκεί ε, επιδιώκουμε να διαπιστώσουμε τις ανάγκες για να αναπτύξουμε τα σωστά προγράμματα για το ανθρώπινο κεφάλαιο. Επίσης, ε, προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε και να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, συνεργαζόμενοι με τους κυβερνητικούς φορείς, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών, ε, στις χώρες ε, που ε, καλύπτουμε. Η ανάπτυξη δυναμικού, το λεγόμενο capacity building, στοχεύει και στη διεύρυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι σε πολλές χώρες που είμαστε παρόντες υπάρχουν διαμάχες, υπάρχουν σειράξεις σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε τοπικό. Ίσως, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο Euronews, στο κανάλι Euronews, παρουσιάστηκε μία ταινία ε, για τις σχέσεις Αρμενίας-Τουρκίας. Η Αναφέρθηκε λοιπόν στην ταινία αυτή το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης, Επαγγελματική Κατάρτισης και είπαν ότι μέσω αυτού του Ιδρύματος μπορούν να κάσουν στο ίδιο τραπέζι ε, αντιμαχόμενες πλευρές για να καταλήξουν σε θετικά αποτελέσματα. Βλέπετε λοιπόν πόσο η επαγγελματική κατάρτιση ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπόρεσαν να συνεργαστούν οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, οι δύο αντίπαλοι και δεν είναι εύκολο να, να τους πείσουμε να συνεργαστούν, αλλά όταν έχει κανείς καλές θετικές πολιτικές που μπορεί να, να, εφαρμοστούν, η, η, η επιτυχία είναι εφικτή. Άλλη πραγματικότητα αρνητική που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η φτώχεια. Η φτώχεια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ε, στη το, πρόγραμμα το εκπαιδευτικό μας επιδιέκουμε την διαφάνεια αλλά και την παροχή ευκαιριών όχι μόνο στους νέους αλλά και στους ενήλικες να, του, να συμμετάσχουν δηλαδή και αυτοί στα προγράμματα κατάρτισης. Ε, επίσης ε, έχουμε, είχαμε αναπτύξει το 2009 προγράμματα ε, ενημέρωσης και ανταλλαγών. Ανταλλαγής πληροφοριών και επισκέψεων. Και όπως είπε και η Διευθύντρια, ε, η κυρία Μπουλγαρέλη, του Ιδρύματος Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης, το 2009 ήταν το έτος διεύρυνσης, ανάπτυξης του ε, πλαισίου επαγγελματικών προσόντων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το πρόγραμμα έχει την μέγιστη υποστήριξη των ε, αδελφών ιδρυμάτων. Ε, συνεργαζόμαστε σε αυτό το πλαίσιο των ευρωπαϊκών ε, προσόντων. Επίσης συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι βρίσκονται στις χώρες που καλύπτουμε η Τράπεζα Ανάπτυξης της Ασίας ε, και πολλοί άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Στόχος μας είναι να επιτύχουν οι χώρες αυτές ε, την αηφόρο ανάπτυξη ε, και την κοινωνική ενσωμάτωση. Το 2009 ο προϋπολογισμός μας ε, ε, ο προϋπολογισμός μας είχε μηδενικό αποτέλεσμα, δηλαδή εάν δεν είχαμε ούτε πλεόνεσμα ούτε έλλειμμα. Τώρα όμως το 2009 όπου δεν είχαμε εξωτερικά προβλήματα, ελπίζουμε να βελτιωθεί η κατάσταση. Οι ελεγκτές που έκαναν τον έλεγχο του 2008-2009, παρόλο που το αποτέλεσμά μας ήταν μηδενικό, ε, βρήκαν κάτι πολύ, μικρο, πολύ πράγματα τα οποία έπρεπε να διορθωθούν, ελάχιστες δηλαδή, ελαχιστότατες παρατυπίες. Το 2010 θα ξεκινήσει η διαδικασία του Τωρίνο, η οποία καλύπτει την επαγγελματική κατάρτιση σε όλες τις χώρες και το 2010 θα μεγιστοποιήσουμε την παρέμβασή μας Όσον αφορά την προσθήκη ε, μέγιστης αξίας στα προγράμματά μας, προστιθέμενης αξίας, ε, τα οποία θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανή βεβαίως και αποτελεσματικά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 2020, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 2020, θέλουμε να διαχειριστούμε σωστά το θέμα της μετανάστευσης για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό που προσφέρει το μεταναστευτικό κεφάλαιο στην Ευρώπη. Αυτό το ζητήσατε από μας και καταγράφουμε όλα τα στοιχεία που περνούν από το Ίδρυμά μας. για να ανταποκριθούμε και στο, στους μεσοπρόθεσμους στόχους του 2013. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τη βοήθειά σας και την υποστήριξή σας ε, για, προς το Ίδρυμά μας. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρουσιάσεις. Έχουμε μερικούς ευρωβουλευτές που ζήτησαν το λόγο για να υποβάλουν ερωτήσεις. Ξεκινούμε πρώτα από την κυρία Ελιζαμπέτ Μοχό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω ε, τους τρεις εκπροσώπους των οργανισμών που μας παρουσίασαν πολύ τεκμηριωμένες εκθέσεις για το έργο τους Ε, γύροντα ε, το ενδιαφέρον τη επιτροπή μας, γιατί είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν όλου αυτά. Χρειαζόμαστε όμως κάποιε επιπλέον διευκρινήσεις και εξηγήσει για τα θέματα των αρμοδιοτήτων. Σας βλέπω ότι έχετε εργαστεί άοκνα για τα ζητήματα που σας απασχολούν και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια διασταύρωση των ιδεών μας και των ανησυχιών μας και ίσως μπορείτε να μας ε, διαφωτίσετε και σε ορισμένε απορίε μα. Έχω λοιπόν μια ερώτηση προς την ε, Διευθύντρια του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, του Ιδρύματος Επαγγελματική Κατάρτισης. Διαπιστώνουμε ότι σήμερα χρειαζόμαστε κάποια κοινά εργαλεία, κάποια κοινά μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να διαμορφώσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο κατάρτισης και εργασίας και να διευκολύνουμε τη κινητικότητα. Παρά τις προσπάθειες όμως, τις προσπάθειες που καταβάλουμε και ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το θέμα του πλαισίου προσόντων, τις πιστώσεις για την κατάρτιση, ε, τα εχέγγυα ποιότητα κτλ. Αυτά τα πραγματευτήκαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία στην Επιτροπή μας. Παρά τις προσπάθειές μας όμως, σήμερα διαπιστώνουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ένας χάρτης κατάρτισης ε, πολύ κατακαιρματισμένος ε, που βρήθη διαφορετικών διπλωμάτων και πτυχίων που δυστυχώς δεν έχουν αντίκρισμα στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει αντιστοιχεία, κάτι που παρεμποδίζει την επαγγελματική κινητικότητα. Το περιεχόμενο ενός επαγγέλματος σε ένα, χάρος, ε, σε ένα κράτος δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του ίδιου επαγγέλματος σε άλλο κράτος. Χρειαζόμαστε λοιπόν εκεί μια καλύτερη, πιο διορατική καθοδήγηση και ίσως ε, ε, να δείξουμε κάποια πυγμή και αποφασιστικότητα και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να διευκρινίσουν ε, την προσφορά της κατάρτισής τους. Χωρίς να επέμβουμε υπερβολικά, χρειάζεται μια τέτοια πίεση, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να διαμορφώσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κατάρτισης και εργασίας. Ερωτώ λοιπόν ποια είναι η γνώμη σας, πώς βλέπετε εσείς αυτές τις εξελίξεις και τι είδου ε, συμβουλές θα μπορούσατε να μας δώσετε. Πάλι προς την ε, Διευθύντρια του ΣΥΤΕΦΟΠ για το θέμα της προσαρμογής των εργαζομένων στην εξέλιξη των θέσεων απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Και εκεί η επιστοποίηση της εμπειρίας, ε, η πρόσβαση στην κατάρτιση για την απόκτηση προσόντων κτλ. είναι θέματα προσφυλή και πάνε πάνω από 10 χρόνια που τα εξετάζουμε αλλά χρειάζονται βαθιές αλλαγές στην ίδια την έννοια της κατάρτισης. Και πριν προσαρμόσουμε τους εργαζόμενους ε, στις εξελίξεις των θέσεων απασχόλης, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την προσαρμογή των ε, εκπαιδευτών, ώστε να εξασφαλίσουν αυτή την επιμόρφωση και τη διαβίου κατάρτιση. Γιατί πολλά λέμε και για πολύ χρόνο συζητούμε αυτά τα θέματα, αλλά δυστυχώ ορατή πρόοδο δεν βλέπουμε. Έχω και μία δεύτερη δέσμη ερωτήσεων προς τον εκπρόσωπο του Eurofound. Διαπιστώνουμε ότι απαιτείται ένας εξυγχρονισμός του χώρου εργασίας μας. Είπατε ότι ο κοινωνικός διάλογος βαίνει καλός. Όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Μήπως και εκεί χρειάζεται ένας εξυγχρονισμός. Ποια είναι τα στοιχεία του εξυγχρονισμού που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις μέσω της κρίσης, γιατί μιλήσαμε για την ελαστικότητα. Τι μπορούν να, να κάνουν επιχειρήσεις σε μια περίοδο κρίσης ε, για να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις απασχόλησης. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τα θέματα αυτά και ένας προβληματισμός που είναι κοινό στα μέλη της Επιτροπής μας είναι ότι επειδή εξετάζουμε τους διάφορους τομείς και τις εξελίξεις τους στην εργασία, ερωτώ, ποιο είναι ο χρόνος απόκρισης για την κατάρτιση και ο χρόνος αντίδρασης για τις αλλαγές στην απασχόληση. Πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την αποτελεσματικότητά μας ό,τι αφορά αυτό το χρόνο αντίδρασης. Γιατί μας μιλήσατε για την αποτελεσματικότητα στις δομές των οργανισμών σας, αλλά πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας. Αυτά τα θέματα με παθιάζουν, γι' αυτό και υποβάλλω τέτοια σώρια ερωτήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την ε, επαγγελματική κατάρτιση. Πώς θα επιταχύνουμε το πέρασμα από το σχολείο στην ενεργό δράση, στην εργασία, γιατί η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει και την κατάρτιση. Πώς όμως μπορούμε να συνδέσουμε άμεσα το σχολείο με την επαγγελματική ζωή. Αναφερθήκατε και στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού πνεύματος ε, στην επαγγελματική κατάρτιση. Θα ήθελα αυτό το πνεύμα να πριτανεύει σε όλες τις φάσεις της κατάρτισης. Γιατί σε περίοδο παγκοσμιοποίησης και κρίσης, όλοι οι νέοι που ολοκληρώνουν μια κατάρτιση θα αντιμετωπίσουν αυτό το επιχειρησιακό πνεύμα. Και όλοι το χρειαζόμαστε. Πώς λοιπόν μπορούμε να επιταχύνουμε την απόκτηση αυτή αυτό και δεν θέλω μόνο πολύ στη συζήτηση, γι' αυτό κάνω χαρακτήρι και περικόπτω τις επόμενες μου ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σέρκας και αν θέλει άλλος κανείς ε, το λόγο για ερωτήσεις. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Σέρκας και μετά θα ξαναδώσω το λόγο σε εμπειρογνωμονούς εκπροσώπους των οργανισμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και εκπρόσωπος του ΕΛΚ και εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά, γιατί αυτό απαιτεί το πρωτόκολλο, η αυρότητα, αλλά και η ειλικρίνη και ο σεβασμός μας προς το έργο που επιτέλεσαν κατά το 2009 οι τρεις οργανισμοί, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία και τις εκθέσεις που μας υπέβαλαν. Εγώ είμαι μάρτυρας για το έργο των δύο οργανισμών, του Μπιλμπάου και του Δουβλίνου. Αλλά και οι άλλοι οργανισμοί επέδειξαν ποιοτικό έργο. Πριν επισέλθω σε συγκεκριμένα ζητήματα, θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση, όχι επικριτική, αλλά αυτοκριτική. Mm. Εμείς, όλοι εμείς που εργαζόμαστε στα κοινοτικά θεσμικά όργανα, καταλήγουμε σε ένα παράδοξο. Βλέπουμε το τεράστιο δυναμικό που έχουμε, ε, κατανόησης, εξήγησης των φαινομένων και ταυτόχρονα έχουμε επιτακτική ανάγκη, τεράστια ανάγκη οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών να μάθουν όλες αυτές τις διαγνώσεις. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να γεφυρώσουμε τις δυνατότητες διάγνωσης που έχουμε και παρατήρησης και των αναγκών. Δυστυχώς δεν μπορούμε να παντρέψουμε αυτά τα δύο σκέλη. Φαίνεται ότι το καθένα ακολουθεί τη δική του πορεία. Είναι σαν να είμαστε ένας κινητήρας άριστα εξοπλισμένος, με απόλυτη λειτουργία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να, να μεταδώσουμε αυτήν την ορμή στις ρόδες, γιατί δεν υπάρχει σωστή διάδραση και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τις πλούσιες εμπειρίες μας στον κόσμο που χρειάζεται αυτή την εμπειρία για να εκμεταλλεύεται την προστιθέμενη αξία. Κάπου λοιπόν κάτι λείπει. Δεν λέω ότι λείπει στου οργανισμού, κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επικοινωνιακή μα πολιτική φταίει. Μπορεί. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει δυσφορία στους πολίτες. Και ήδη κάνουμε πολλά, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο, να βελτιώσουμε στο μέλλον την επικοινωνιακή μας πολιτική. Κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να βελτιώσουμε και τον τρόπο επαφής μας ε, με την πραγματικότητα. Γιατί όταν έχουμε άδειες εκκλησίες ε, ε, και ενορίες, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ε, ιερέων. Αυτούς που μένουν ε, με σταυρωμένα χέρια στι άδειες εκκλησίες και αυτούς που βγαίνουν και προσπαθούν να προσιλητήσουν ή να ξαναφέρουν τον κόσμο το πίμνιό του στην εκκλησία. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς, ή να υιοθετήσουμε παθητικό ρόλο ή ενεργητικό. Να βγούμε στον δρόμο, να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες, στις πιο απρόσμενες ε, περιοχές και χώρους, αλλά να μην μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, να ρωτήσουμε τον κόσμο να έρθουμε σε επαφή άμεση μαζί του. Και αυτή είναι μια υπόδειξη προς τις οργανισμούς. Αν περιμένετε οι ευρωβουλευτές να έρθουν σε εσά, να σας πω, οι ευρωβουλευτές έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας. Έχουμε τόσο πολλά να κάνουμε που δεν πηγαίνουμε καν στην ενορία μας να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία. Δηλαδή δεν ερχόμαστε στις συνεδριάσεις ε, των επιτροπών. Αυτό είναι ένα θέαμα που δικαιολογείται σήμερα. Αλλά όταν έρθετε εσείς ε, και μας ενημερώσετε θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα γιατί σας χρειαζόμαστε. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα από, την, ε, από τον οργανισμό του Βελβάο με εντυπωσίασε η επίσκεψη που πραγματοποίησα εκεί και μάλιστα ρώτησα και το θέμα στον Ισπανό Υπουργό και μου είπε ότι επιτέλους διευθετούνται τελικά προβλήματα. Πάντως εγώ εντυπωσιάστηκα από το έργο του οργανισμού του Μπιλμπάου και εντυπωσιάστηκα από τη μετριοφροσύνη σας σε σχέση με το, το ποιοτικό έργο που επιτελείται στο Βιλμπάο. Και θα ήθελα κύριε Τακάλα, με τη φιλία που τρέφω απέναντι σας και το σεβασμό, να σας πω ότι μετά από το προβληματισμό σας για την αξιοπρεπή εργασία και τα θέματα της στρατηγικής του 2020, θέματα που αποτελούν ουσιαστικά ακρογωνία ηλίθους της μελλοντικής μας Ευρώπης. Θα ήθελα και εμείς είχαμε παρόμοιες ανησυχίες και να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμός μεταξύ των οργανισμών. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν ή εσείς να μας δώσετε κάποιο έγγραφο, όχι μόνο στην Επιτροπή, στο ίδιο το Κοινοβούλιο, όταν έχουμε στοιχεία από τη ΔΟΕ, όταν έχετε εσείς στοιχεία από τη ΔΟΕ, χρήσιμες πληροφορίες, να τις στέλνετε εσείς στους Ευρωβουλευτές, για να ενημερωθούμε για την πραγματικότητα. Μπορείτε να μας υποδείξετε ή να μας προτείνετε κάποιες πρωτοβουλίες που θα χρειαστούν να αναλάβουμε για να ικανοποιήσουμε αυτές τις κοινέ μας ανησυχίες. Και έτσι θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε όχι μόνο τις ανησυχίες αλλά και τα προγράμματά μας, όχι μόνο του Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου. Και όταν βλέπετε ότι υπάρχει κάτι στο πολιτικό μας πρόγραμμα, ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να μας στέλνετε πληροφορίες, συμβουλές, προτάσεις. Αυτό είναι εύκολο και θα σας είναι ευγνώμονες και οι συγητές των διαφόρων εκθέσεων και οι επιτροπές. Και εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μα ώστε να μην πηγαίνει ο Μωάμεθ στο βουνό, αλλά το βουνό στο Μωάμεθ θα έρχεστε εσείς σε εμά. Και έτσι θα μα βοηθήσετε και στο έργο μα. Γιατί εκτό από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, προσέξτε λίγο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσπαθήστε να ευθυγραμμιστείτε κάπω και με το δικό μα πολιτικό έργο. Και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, προ τον κύριο Καρπίνα. Θα ήθελα να πω ότι συγχαρητήρια γιατί είναι καταπληκτικό το έργο του οργανισμού και υπάρχει το γραφείο τη Βρυξέλλες Έχω πολύ αγαστή συνεργασία μαζί σας και θα συνεχίσω να έχουμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του Eurofound. Χρειαζόμαστε και τη δικιά σας βοήθεια και σας παροτρύνω να μην είστε τόσο άτολμοι και εσείς να αναλάβετε πρωτοβουλία, να μας στείλετε έγγραφα. Μην περιορίζετε μόνο στα ακαδημαϊκά και θεωρητικά ζητήματα. Τολμήστε, όπως κάνει ο οργανισμός του Μπιλμπάου. Σήμερα το απόγευμα θα εξετάσουμε θέματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Ε, για αυτούς που πραγματοποιούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Στείλτε μας πληροφορίες σχετικά. Γιατί δεν έχουμε τέτοια υποστήριξη από, τις, από τους οργανισμούς. Πώς επηρεάζει το θέμα της ασφάλειας, ε, ε, το, το ωράριο εργασίας και ατέρμονες ώρες εργασίας. Ε, υπάρχει φοβερή τεχνογνωσία στις, στους οργανισμούς σας, γι' αυτό τη χρειαζόμαστε. Κυρία Βουλγαρέλη, θα ήθελα να μου στείλετε παρακαλώ τη σύνοψη αυτού του, αυτής της εξωτερικής αξιολόγησης και τους δείκτες των αποτελεσμάτων. Γιατί θα, θα ήθελα του χρόνου να μπορώ να μιλήσω ε, πιο ενημερωμένος για το ΣΕΔΕΦΟΠ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Σερεβάν για το έργο της και να της ευχηθώ επίσης καλή επιτυχία. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις που προσεγγίζουν ε, τις δικές σας. Προσπαθούμε να βρούμε ένα τρόπο να συνεργαστούμε περισσότερο μαζί σας. Ορισμένοι από εσά συνεργάζεστε μαζί μας σε προσωπικό επίπεδο. Ε, ορισμένες φορές λείπουν πολλοί ευρωβουλευτές. Γι' αυτό ε, προσπαθώ να βρω έναν καλύτερο τρόπο συνεργασίας. Ίσως ε, μικρότερης κλίμακας με λιγότερους συμμετέχοντες ή συνεργασία πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, σε διαφορετικούς τομείς. Θα ε, ήθελα λοιπόν να ξέρω, επειδή μας αναφέρετε τις επιτυχίες σας τα τελευταία χρόνια, θα ήθελα λοιπόν να ξέρω σε όσους δεν μας ανέφεραν τα καλύτερά τους επιτεύγματα, ε, τι θεωρούν ότι ήταν η μεγαλύτερη τους επιτυχία το 2009. Ε, ίσως ε, η, ενίσχυση, η συμβολή στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συμβολή στις εργασίες της Κομισιόν. Για ποιο λοιπόν επίτευγμα είσαστε υπερήφανοι, ποιο ήταν το καλύτερο, η μεγαλύτερη σας επιτυχία και ε, θα αρχίσω επειδή είμαστε και πιεσμένοι από χρόνο, θέλουμε να τελειώσουμε στις 5 παρατέταρτο, ε, θα ήθελα να, να αρχίσω με τον κύριο Τάκαλα. Thank you very much. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω από την τελευταία σας ερώτηση. Ποια ήταν η μεγαλύτερη μας επιτυχία. Πιστεύω ότι ήταν η εκστρατεία μας για την αξιολόγηση κινδύνων, την αξιολόγηση του ρίσκου, η οποία έφτασε σε περισσότερο από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους εργαζόμενους. Και συνεργαστήκαμε και με ένα τεράστιο αριθμό αρμοδίων φορέων και ιδρυμάτων, 65, ε, ε, Είμαστε λοιπόν πολύ ευτυχής για αυτή την επιτυχία και ένα άλλο που μας καθιστά πάρα πολύ ευτυχής είναι η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, με το Κοινοβούλιο. Η Ισπανική Προεδρία τώρα έχει πάρα πολλά προγράμματα τα οποία θίγουν τις δικές μας αρμοδιότητες, ε, ε, άπτονται των δικών μας αρμοδιοτήτων και γι' αυτό πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα είναι ακόμα πιο στενή και επιτυχημένη. Ε, όπως ε, είπε ο κύριος Σέρκας, ε, υπάρχει μεγάλη αλληλοϊποστήριξη των εργασιών μας και τρίτον, προσπαθούμε να βρούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να καλύψουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020. Όπως σας είπα, έχοντας τη μεγάλη εμπειρία της μακροχρόνιας εργασίας στη Γενέβη, στο Διεθνή, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ε, ε, μπορώ να, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα ακολουθούμε διαφορετικούς δρόμους. Θα ακολουθούμε παράλληλους δρόμους και ε, την ίδια κατεύθυνση. αυτό το οποίο με ευχαριστεί ιδιαίτερα είναι όταν βρίσκουμε εφαρμογές που αφορούν συγκεκριμένα το χώρο εργασίας, διότι εκεί παρουσιάζονται τα πραγματικά προβλήματα. Στο χώρο εργασίας παρουσιάζονται τα προβλήματα και εκεί πρέπει να βρούμε και τις λύσεις. Το δίκτυό μας είναι εκτεταμένο, το δίκτυο συνεργασίας. Ακόμα και οι κυβερνήσεις βεβαίως είναι εργοδότες και αυτό το εκτεταμένο δίκτυο μας δίνει τεράστια εμπειρία και γνώση. Το, η ιστοσελίδα μας η οποία μπορεί να, να παρουσιαστεί σε 22 διαφορετικές γλώσσες, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή σε 22 διαφορετικές γλώσσες, είναι επίσης και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό πιστεύω ότι είναι μια ε, επιτυχία μας η δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας, σαν πηγή πληροφοριών. Ε, η κυρία Βουλγαρέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω να απαντήσω σύμφωνα. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το κύριο επίτευγμά μας ε, για το 2009. Νομίζω ότι ήταν ακριβώς το ότι καταφέραμε να δώσουμε ε, στοιχεία αποδεικτικά, μαρτυρίες για τις βέλτιστες πρακτικές. Πρόκειται για θέμα το οποίο ήταν στην ημερησία διάταξη πέρσι και είναι και φέτος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη-μέλη και ε, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κυρίως το Συμβούλιο και οι Κομισιόν ε, χρησιμοποιούν τις αναλύσεις μας έτσι ώστε να ε, δώσουν μορφή σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και η Τσεχική Προεδρία όπως και η Σουηδική Προεδρία προσέφυγε στις υπηρεσίες μας κατά αυτή την έννοια. Θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ με τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που μου ε, ο κύριος Βουλευτής. Ναι, ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να προσαρμόσουμε ε, το περιεχόμενο των διπλωμάτων ε, και της κατάρτισης. Αναφερθήκατε στα εργαλεία τα οποία τα γνωρίζετε πολύ καλά. Πρόκειται για εργαλεία τα οποία πλέον είναι ευρωπαϊκού επίπεδου έτσι ώστε να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα. Όμως ε, το η πραγματική δύναμη του εργαλείου είναι κυρίως παραδειγματική. Εξηγούμε από το input μέχρι το output της γνώσης και της εκμάθησης η διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και έχουμε τώρα μία μετατόπιση από τις παραδοσιακές μορφές διπλωμάτων, πτυχίων ε, που αυτή τη στιγμή υπολογίζονται ως input, δηλαδή ως χρόνια σπουδών και ένα, μια μετατόπιση από το input στο output, δηλαδή τι έχει μάθει κανείς στο, κατά το πέρασε της διαδικασίας ε, μάθησης. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ οι επίσημες γνώσεις που ε, παίρνει κανείς στη διάρκεια της επίσημης διαδρομής σπουδών, αλλά κάθε είδους γνώση ή δεξιότητα την οποία έχει επιτόπου ενδεχομένως και λόγω δουλειάς αποκτήσει. Νομίζω ότι διαπιστώνουμε μικρές επαναστάσεις όσον αφορά ε, την ε, μάθηση βλέπουμε ότι σιγά σιγά τροποποιείται ε, και η επαγγελματική κατάρτιση αλλά και η εκμάθηση στα πανεπιστήμια σε περιοριστικό επίπεδο τροποποιείται λέγω και μετατίθεται σιγά σιγά από την σημασία στο input ε, στην σημασία στο output. Και ε, κατά την αντίληψη αυτή είναι πολύ σημαντικό να δούμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ε, προσαρμοστικότητα. Πολύ δουλειά έχει γίνει, ιδίως από το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι δεξιότητες, αλλά κυρίως για να γίνουν κατανοητές οι αποδόσεις ή ε, επιδόσεις που χρειάζονται ε, επιτόπου στις ε, θέσεις εργασίας. Επομένως, υπάρχει μετατόπιση προς, τις, προς την απόδοση, προς τις συγκεκριμένες επιδόσεις, αλλά και προς αυτήν την εγκάρσια προσπάθεια αντιμετώπισης που αφορά ας πούμε την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσης, την ικανότητα λύσης προβλημάτων ε, με ταχύτητα κτλ. Αλλάζει λοιπόν το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας, αλλάζουν οι απαιτήσει ε, οι εργασιακές και επομένως αυτό ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος παροχής, εκπαίδευσης, γνώσης ή κατάρτισης. Πολλά μπορούμε να πούμε γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο. Ε, πάντως, ε, τελειώνοντας να πω ότι τον Μάρτιο θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος τα θέματα αυτά. Όσον αφορά το, την επικοινωνία, είναι γεγονός ότι το Σέντεφοβ είναι λίγο ντροπαλό στέλνουμε κάποιες briefing notes, κάποια ενημερωτικά ε, σημειώματα, τα οποία είναι πάντα πάρα πολύ σύντομα, είναι επιγραμματικά. είναι γεγονός ότι θα θέλουμε, θα θέλουμε να βελτιώσουμε την ροή επικοινωνίας και να σταματήσουμε να είμαστε τόσο ντροπαλοί. Σας ευχαριστώ κύριο Σκάρπινεν από Σας ευχαριστώ. κρίνοντας από τις αδελφές υπηρεσίες, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά επιτεύγματα αξιομνημόνευτα και εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ δύο-τρία. Για παράδειγμα, εκτεταμένη χρήση των δεδομένων παρακολούθησης. Είναι ο ταχύτερος τρόπος παρακολούθησης του τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Γιατί είχαμε στενέ επαφέ με τον Επίτροπο Σπίτλα, από όλου του Ευρωβουλευτέ και πολλέ οργανώσει που χρειάζονται τα στοιχεία μα, τα δεδομένα μα ταχύτατα. Και αυτό ήταν σημαντικό επίτευγμα του Eurofound. Πολλά βασικά έγγραφα, σημαντικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπουν στον οργανισμό μας. Υπάρχουν πάνω από 80 ε, μνήες έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό επίτευγμα. Είμαστε σημείο αναφορά. Επίσης, ε, έχουμε πολλές εκθέσεις ε, ακριβεί ε, που ανταποκρίνονται στι ανάγκε πληροφόρηση πολλών ευρωπαϊκών οργανώσεων και θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένων και του Κοινοβουλίου. Επίσης, συμμετέχουμε τακτικά σε πολύ σημαντικέ ομάδε εργασία που διαμορφώνουν ουσιαστικά το μέλλον της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτά αρκούν. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σέριαν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τις δικές σας ερωτήσεις που νομίζω ήταν προς εμένα απευθείας. Πώς θα βελτιωθεί η επικοινωνία. Καλό θα ήταν στο πρόγραμμα εργασίας να περιλαμβάνουμε και την εξωτερική διάσταση όπου χρειάζεται. Επίσης, ε, σε ποιες θεματικές ενότητες χρειάζεται τη δική μας ε, σύμβολη και συνεργασία. Επίσης, έχετε και τους ε, διορισμένους σας εμπειρογνώμονες και αυτοί με τις προτάσεις τους μπορούν να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που μπορούν να, να περιλαμβάνονται και στο δικό σας πρόγραμμα και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020. Βέβαια, ξέρουμε ότι έχετε φόρτο εργασίας και προσπαθείτε να το διαχειριστείτε όσο καλύτερα μπορείτε. Πάντως είμαστε στη διάθεσή σας. Είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε ό,τι πληροφορίες χρειάζεστε. Το βασικό επίτευγμα για το 2009 και πόσο περήφανοι αισθανόμαστε. Αυτό είναι το πιο δύσκολο να κρίνει κανεί. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαίνεται ότι η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για όλες τις προγραμματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες δωρητών προσκληθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμβάλλουμε στη συζήτηση. Αυτό δείχνει πόσο ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπιστεύεται την εμπειρογνωμοσύνη μας και το, την τεχνογνωσία μας. Έχουμε στενές συνεργασίες με τις χώρες εταίρους, δίνουμε έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία και αυτός ο διακρατικός και διαπεριφερειακός διάλογος είναι πολύ σημαντικός, γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Είμαι στη διάθεσή σας να σας ενημερώνω τακτικά. Αυτό πάντως ε, που εμπνέει τις χώρες ε, εταίρους είναι τα διάφορα έγγραφα, επίσημα έγγραφα των τριώθεσμικών οργάνων. Οπότε η στρατηγική του 2020 θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση. Γιατί χρειαζόμαστε ανώτατη εκπαίδευση, αλλά πώς θα συμβάλλει η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση στην ανάκαμψη από την κρίση. Νομίζω ότι έχει νόημα να συμπεριληφθεί και αυτές τις προτεραιότητες της στρατηγικής του 2020. Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνική ένταξη. Το είπα και στην παρουσίασή μου. Σε όλες αυτές τις χώρες το θέμα της κοινωνικής ένταξης είναι κέριο, έχει νευραλγική σημασία. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ε, ενδιαφέρει όλους η κοινωνική ένταξη και ίσως η στρατηγική του 2020 θα δείξει τη την τεράστια οικονομική προσπάθεια που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και ο πιο γενναιόδωρος δωρητής. Έτσι θα δώσετε και σε εμά την ευκαιρία να εμπλακούμε σε αυτή τη διαδικασία και στην επόμενη παρουσίαση που θα σας αναφέρω τα βασικά μας επιτεύγματα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Τώρα η μετάβαση από το σχολείο στη δουλειά και το επιχειρηματικό πνεύμα. Αυτό στις τρίτες χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι κέρια σημασία. Η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Όταν λέμε σχολείο, εννοούμε γενικά τους παρόχους ε, επιμόρφωσης και κατάρτισης, ακόμη και διαβίου κατάρτισης και επαγγελματική κατάρτισης. Πώς την ενθαρρύνουμε με το διάλογο μεταξύ των δύο κόσμων, της επαγγελματικής κατάρτισης και του επιχειρηματικού κόσμου. Σε πολλές χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, δυστυχώς αυτοί οι δύο κόσμοι, αυτοί οι δύο κύκλοι είναι ξεχωριστοί και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Γι' αυτό το Δεκέμβριο οργανώσαμε μια τέτοια συνδιάσκεψη που κάθισαν πρόσωποι των δύο κύκλων στο ίδιο τραπέζι. Και φαίνεται αυτό και στα χαρτιά που σας δώσαμε, Προσπαθούμε να καταρτήσουμε μια λεπτομεριακή μελέτη για το πώς θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε αυτό το διάλογο, τι ενάψματα θα πρέπει να δώσουμε και θα προτείνουμε στις χώρες εταίρους κάποιες πρωτοβουλίες, είτε στον προγραμματισμό είτε στις δραστηριότητες ε, του κέντρου μας, για να κάνουμε πραγματικότητα αυτή τη μετάβαση από το σχολείο, από τις σπουδέ στην εργασία. Το 2009 το χαρακτηρίσαμε την αναγέννηση της κατάρτισης και της μαθητείας. Χρειαζόμαστε συνεργασία για την επαγγελματική κατάρτιση, για να γίνονται στα μαθητείες στην επιχείρηση, στις επιχειρήσεις, να μην είναι ε, απομονωμένοι κόσμοι τα πανεπιστήμια από τις επιχειρήσεις, να μην είναι σε έναν για άλλο πύργο απομονωμένη από την πραγματικότητα της δουλειάς. Επίσης, σημαντικό είναι και το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της καθοδήγησης. Γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη ε, διαφορά και δυστυχώς δεν ταιριάζουν ε, η ζήτηση στην εργασία και η καθοδήγηση στην, στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Θα πρέπει να προσαρμοστούν οι ανάγκες στην προσφορά. Δεν θα πρέπει οι δύο κόσμοι αυτοί να είναι ξεχωριστή. Τώρα, για να ενισχυθεί το επιχειρηματικό πνεύμα, το πιο σημαντικό μήνυμα προς χώρες εταίρους είναι να τους πούμε και να, το, να κατανοήσουν ότι η επιχειρηματικότητα για το επιχειρηματικό πνεύμα δεν σημαίνει μόνο η ίδρυση μιας επιχείρησης. Σημαίνει και ένα προσόν, μια δεξιότητα που θα πρέπει να ξεκινάει από την πρώιμη διαπαιδαγώγηση, από την παιδική ηλικία. Να λαμβάνουν υπόψη ανάγκες του, της κάθε ομάδας και να μην καθοδηγούμαστε μόνο από ένα εμποροκρατικό πνεύμα. Πάντως οι χώρες εταίροι με τις οποίες συνεργαζόμαστε, που είναι πολλές, αντιλαμβάνονται αυτή την ανάγκη. Και με τη βοήθεια των βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών, συνεργαζόμαστε μαζί τους για την διάδοση αυτών των βέλτιστων πρακτικών. Γιατί η επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα δεν σημαίνει κατά ανάγκη, και το είπε και αυτό και η διευθύντρια του ΣΕΤΕΦΟΠ, δεν σημαίνει μόνο εμπορικό πνεύμα. Θα πρέπει να διευρύνουμε το διάλογο μεταξύ των χωρών, μερών και των, των χωρών μελών και των uh, χωρών εταίρων, των τρίτων χωρών. Δεν ξέρω αν απάντησα σε ερωτήσει είμαι στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντας ε, στο πάνελ. Ρώτησα ποια είναι τα μεγαλύτερη σας επιδέγματα, διότι είσαστε τόσο μετριοπαθείς που πιστεύω ότι σήμερα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να γνωρίσουν όλοι τι, έχετε καταφέρει και τι μπορείτε να κάνετε. Δεν έχουμε πολύ συχνά την ευκαιρία να σας ακούσουμε ομαδικά. Σας ευχαριστώ όλους για την εξαιρετική σας ενημέρωση και ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονές μας που ήρθαν σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, η επόμενη μας ε, γνωμοδότηση είναι η οργάνωση του χρόνου εργασίας ε, των εκτελούντων κινητές δραστηριότητε οδικών μεταφορών. Edith Bauer. We'll uh, Να περιμένουμε δύο-τρία λεπτά ώσπου να τακτοποιηθούμε. Those Παρακαλώ, όσοι φεύγετε από την αίθουσα, αποχωρήστε σύντομα για να συνεχίσουμε. Θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Σας παρακαλώ, αποχωρήστε γρήγορα από την αίθουσα για να δώσω το λόγο στην κυρία Μπάουερ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αρχίσω με αυτό το πολύ ε, ενδιαφέρον, αντιφατικό και ενδιαφέρον θέμα. Θα μιλήσω ε, ουγγρικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην ουσία πρόκειται για μια μικρή αλλαγή, πολύ μικρή αλλαγή στην νομοθεσία, για την οποία πολύ μικρή αλλαγή όμως είχαμε ατελείωτες συζητήσεις. Και σας εξηγώ γιατί όλοι έχουν τελείως διαφορετικές ιδέες σχετικά με το τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μικρή αλλαγή. Μικρή αλλαγή λοιπόν με πολύ, με πολύ μεγάλο σημαντικό αντίκτυπο ε, όσον αφορά τους εργαζόμενους στον ε, τομέα που μας ενδιαφέρει. Πρόκειται για τρεις ώρες σχετικά με τους εκτελούντες κινητές δραστηριότητες που δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση. Πρέπει να μιλήσουμε για τις τρεις ε, ώρες, πρέπει να μιλήσουμε για χρόνο οδήγησης, αλλά βεβαίως πρέπει να μιλήσουμε και για ε, κοινωνικά θέματα, πρέπει να μιλήσουμε και για ασφάλεια στους δρόμους μας να σας πω ότι αυτή η αλλαγή νομοθεσίας δεν αφορά την, και δεν θα έχει αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια. Εάν θέλει κανείς να μιλήσει για οδική ασφάλεια θα πρέπει να το κάνει στα πλαίσια άλλης νομοθεσίας. Εδώ γίνεται λόγος μονάχα για τους εκτελούντες κινητές δραστηριότητες, για αυτούς τους εργαζόμενους δηλαδή. Υπάρχει ένα κείμενο του 2002 που αναφέρεται στην οδική ασφάλεια. Έχουμε επίσης Έχουμε και την 561 που μιλάει για την οδική ασφάλεια και επίσης την 1071 που αναφέρεται στην οδική ασφάλεια επίσης. Αυτά τα τρία κείμενα τα οποία μόλις ανέφερα αναφέρονται στις ε, συνθήκες που πρέπει να καλύπτονται από τα φορτηγά ή ε, τα άλλα οχήματα τα οποία εκτελούν οδικές μεταφορές. Οτιδήποτε άλλο θα καλυφθεί αλλού. Όσον αφορά τώρα το κοινωνικό dumping, όντως και αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να μας απασχολήσει σε άλλο νομοθετικό πλαίσιο. Δεν θέλω να θεωρήσουν οι συνάδελφοι ότι είμαι υπέρ του κοινωνικού ντάμπινγκ. Δεν ισχύει αυτό. Όμως λέγω ότι θα πρέπει να γίνει αναφορά στο κοινωνικό ντάμπινγκ αλλού και όχι εδώ. Ας δούμε τώρα το ίδιο το κείμενο επανειλημμένα συζητήσαμε και είχαμε μάλιστα πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει για το κείμενο αυτό. Και εγώ προσπάθησα κάθε φορά να εξεύρω ε, κάποιο συμβιβασμό. Πιστέψτε με, σας μιλώ ειλικρινά. Αλλά ήθελα πάντα εφικτές συμβιβαστικέ λύσεις. Υπάρχει πρώτα το θέμα των ψεύδο αυτοαπασχολούμενων. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά και το επαναλαμβάνω απλώς, οι ψεύδο αυτοαπασχολούμενοι δεν αφορούν μονάχα τους μετακινούμενους εργαζομένους, δεν αφορούν δηλαδή μονάχα αυτόν τον τομέα. Ε, ψεύδο αυτοαπασχολούμενοι υπάρχουν σε κάθε ε, κλάδο της οικονομίας. Ε, ζητώ λοιπόν να τροποποιηθούν οι αιτιολογικές σκέψεις ελαφρά και να πούμε ότι το φαινόμενο των ψεύδο αυτοαπασχολουμένων αφορά πολλούς κλάδους. Υπάρχουν πολλές χώρες όπου η φορολογική νομοθεσία είναι τόσο αποτελεσματική που δεν, έχουν, ε, που δεν αφήνονται περιθώρια για, για ε, Πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν στις άλλες περιπτώσεις να καταργήσουμε το φαινόμενο των ψευδοαυτοαποσχολούμενων. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι αυτή, ε, το το πρόβλημα δεν υπάρχει μονάχα στους μετακινούμενους εργαζόμενους, αλλά και σε κάθε άλλο τομέα της οικονομίας. Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα όσον αφορά τα οχήματα οχήματα ε, μικρότερα των 3,5 τόνων, γιατί στα οχήματα αυτά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να καλυφθούν. Όμως νομίζω ότι όλοι οι παριστάμενοι γνωρίζουν ότι η οδηγία για τον χρόνο εργασίας αφορά και τους οδηγούς ε, ε, φορτηγών λιγότερων των 3,5 τόνων. και επομένως θα πρέπει ο χρόνος οδήγησης να αφορά όλα τα οχήματα και όχι μονάχα τα, βαρύτερα, τα οχήματα που είναι βαρύτερα από 3,5 τόνους. Έχουμε λοιπόν και νομοθετήματα τα οποία αφορούν ε, τα ε, οχήματα που ζυγίζουν λιγότερο από 3,5 τόνους. Θα ήθελα τώρα να έχω και την άποψη της Επιτροπής, γιατί δεν ξέρω ακριβώς ε, ποιες είναι οι αποκλήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά τα φορτηγά που είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα των 3,5 τόνων. Στην οδηγία 561 γίνεται αναφορά ε, σε, ε, ψηφιακούς ταχογράφους και εκεί γίνεται διαφοροποίηση ε, στα φορτηγά που είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα των 3,5 τόνων. Επόμενο ζήτημα. Να δούμε εάν το πεδίο εφαρμογής θα καλύψει τους αυτοαπασχολούμενους και τους ψευδοαυτοαπασχολούμενους. Εάν θέλετε τη δικιά μου γνώμη, εάν θέλετε δηλαδή τον τρόπο που βλέπω εγώ τα πράγματα, μπορώ να σας πω το εξής. Στις χώρες όπου υπάρχουν προϋποθέσεις για τον εξορθολογισμό της κατάστασης αυτής μπορούμε να εφαρμόσουμε και την ε, οδηγία για τους αυτοαπασχολούμενους. Νομίζω όμως ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό σε κοινοτικό επίπεδο. Και θα ήθελα να επαναλάβω και κάτι το οποίο επανειλημμένα έχω πει. από τη στιγμή που ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, είναι τμήμα της συνθήκης της Λισαβόνας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ε, μια οροφή όσον αφορά τις ώρες απασχόλησης για τους εργαζόμενους, όμως δεν μπορούμε να καθορίσουμε ένα τέτοιο ε, όριο για τους αυτοαπασχολούμενους. Θα είναι γελίο, λέει ο Μιλήτρια, και θα ήταν και ε, αντιπαραγωγικό. Και, εν πάση περιπτώσει, το λέω με την έννοια ότι δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι η οδηγία για την ε, απαγόρευση του καπνίσματος είναι περίπου το ίδιο πράγμα, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ε, παραλληλισμούς ε, και συγκρίσεις ανάμεσα στο κάπνισμα και τους μετακινούμενους εργαζόμενους πιστεύω ότι ε, τα έχω ξαναπεί αυτά και ελπίζω ότι οι συμβιβασμοί στους οποίους έχω καταλήξει θα γίνουν αποδεκτοί από όλους και θα μας επιτρέψουν επίσης να επιτύχουμε τους στόχους μας και επομένως να δημιουργήσουμε ένα κείμενο το οποίο θα είναι αποδεκτό από όλους. Α, νο, πρέπει επίσης να μιλήσουμε για την νυχτερινή εργασία. Και νομίζω ότι η πιο έξυπνη λύση θα ήταν η εξής. Κάθε κράτος μέλος να μπορεί να καθορίσει την νυχτερινή χρονική περίοδο. Ε, χθες στην Επιτροπή Μεταφορών μας είπε κάποιος ότι δεν δει ο ήλιος την ίδια ώρα στην Φιλανδία και στην Ισπανία. Επίσης ότι στην ε, Ισπανία ή στην Πορτογαλία ας πούμε δεν διπνούν την ίδια ώρα με την οποία διπνούν στην Ουγγαρία. Ε, ας πούμε στο εστιατόριο ένας Πορτογάλος μπορεί να πάει να φάει ανέτος στις 9.30 ε, ενώ, ενώ στην Ουγγαρία 9.30 έχει κλείσει πλέον η κουζίνα στα περισσότερα εστιατόρια. Επομένως θα πρέπει να καθορίσουμε τι εννοούμε ε, νύχτα και νυχτερινή χρονική περίοδο. Και πραγματικά μπορούμε, είναι λογικό δηλαδή να κάνουμε τέτοιου είδους τροποποίησεις όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία. Νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να βρούμε ε, τρόπους, ε, απαραίτητες ε, ρήτρε και νομίζω ότι με τις προτάσεις μου ίσως θα μπορέσετε να συμφωνήσετε. Έχω ένα αίτημα να διατυπώσω. Βοηθήστε μας να κρατήσουμε την ισορροπία αυτού του κειμένου. εάν διατηρήσουμε τους αυτοαπασχολούμενους στο, πλαίσιο της, στο πεδίο της οδηγίας αυτής, εάν οι έλεγχοι αφορούν μονάχα 4% των αυτοαπασχολούμενων, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πολύ ε, σημαντικό κόστος, περισσότερο από το κόστος του ίδιου του ταξιδιού που κάνει το Κοινοβούλιο από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο. Επομένως καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να δεχτείτε τις προτάσεις που έχω κάνει σχετικά με το κείμενο αυτό. Γνωρίζω βεβαίω ότι υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία μπορούν να αποσαφινιστούν και να βελτιωθούν στο κείμενο αυτό. Και εγώ ίδια θα υποβάλω τροπολογίες άλλωστε. Εν πάση περιπτώσει, επίσης έχω λάβει γνωμοδότηση από την ε, Βρετανική κυβέρνηση που μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Μου έμαθε ας πούμε ότι η γνώμη που μπορεί να έχει κάποιος εδώ για την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, μπορεί να διαφέρει από την πραγματικότητα. Ε, γιατί διαπιστώνουμε βάσει της γνωμοδότησης της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ότι ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμπεριλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι σε αυτές τις διατάξεις, ενώ εμείς εδώ είχαμε την αίσθηση ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ. Κύριο Σέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να, να πω στους συναδέλφους ότι δεν είμαστε σαν τους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα. Υπήρχε κόσμος και πριν την έκθεση αυτή. Και είχαμε μακρά παράδοση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκθέσεων για το ωράριο εργασία, για εργαζόμενους που εκτελούν κινητές δραστηριότητες στις οδικές μεταφορές. Και μην ξεχνούμε και τον ε, Ευρωβουλευτή Στίβεν Χιούς που πολλοί πολυάριθμες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σχολίασε και την αρχική οδηγία του 2002. Σήμερα τον αντικαθιστώ γιατί ασθενεί ο κύριος Χιούς, γι' αυτό ε, τον αναπληρώνω εγώ. Αλλά πιστεύω ότι θα πω παρόμοια πράγματα με αυτόν σε μια ίστατη προσπάθεια να μεταπίσω την κυρία Μπάουερ και να ασχοληθώ με ορισμένα πράγματα που είναι ουσιώδη για την οδηγία αυτή. Η κυρία Μπάουερ είπε στο τέλος ότι επιδιώκει ένα συνενετικό κείμενο. Το έγγραφο που έχουμε, η έκθεση αυτή, όχι μόνο δεν είναι συνενετική, αλλά είναι το αντίθετο. Όχι της γνώμης ορισμένων ομάδων, αλλά έρχεται σε αντίφαση με την ίδια τη γνώμη τη δική τη ομάδα κατά τη συζήτηση τη αρχική οδηγία. Αν διαβάσετε, συνάδελφοι, τον τίτλο ε, του νομικού αυτού εργαλείου που έχουμε, είναι «Αναθεώρηση τη αρχική οδηγία του 2002». Δηλαδή, στην οδηγία αυτή περιληφθήκαν οι αυτοαπασχόλου μέλη. Τώρα προσπαθούμε να τους απαλείψουμε, να καταργήσουμε αυτή τη μνήμα. Αν οι αυτοαπασχολούμενοι περιλήφθηκαν το 2002, αυτό έγινε γιατί σύσσωμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμη και η παράταξη της κυρίας Μπάου, είχε συμφωνήσει το 2002 να συμπεριλάβει τους αυτοαπασχολούμενους. Και το 90% των μελών του Συμβουλίου, με εξαίρεση την Ισπανία και τη Φιλανδία, η πλειοψηφία του Συμβουλίου ήταν υπέρ της συμπερίληψης των αυτοαπασχολούμενων. Και η ίδια συνένεση υπήρχε και στην ε, Εκτελεστική Επιτροπή και σε όλες τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς το 2002 καταλήξαμε στη συνένεση αυτή, κατά πάσα πιθανότητα, επειδή οι ερωτήσεις που μας προβλημάτισαν τότε ήταν διαφορετικές από αυτές που θέτει η κυρία Μπάουερ, γι' αυτό και η απάντηση ήταν διαφορετική. Τότε σκεφτήκαμε ο χρόνος εργασίας των οδηγών σχετίζεται με την οδική ασφάλεια και με την ασφάλεια των ίδιων των οδηγών, αλλά και των πολιτών που επίσης οδηγούν στις αυτοκινητοδρόμους. Αυτή ήταν η ερώτηση που είχαμε θέσει τότε. Και εμείς και οι ομοειδεάτες σας, κυρία Μπάουερ, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι για να λάβουμε υπόψη την οδική ασφάλεια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κόποση των οδηγών, που δεν σχετίζεται άμεσα μόνο με τις ώρες εργασίας. Γιατί αν ο οδηγός πριν την οδήγηση έχει και χειρονακτική εργασία, ήδη με το που ξεκινάει να οδηγεί, είναι πτώμα ο άνθρωπος. Θα πρέπει να συνδυάσουμε λοιπόν την οδήγηση με την ε, σωματική εργασία που γίνεται εκτός της οδήγησης, για να μετρήσουμε την κόποση του εργαζομένου. Η κυρία Μπάουερ μας είπε ότι καλύτερα να μην συζητήσουμε θέματα οδικής ασφάλειας. Δεν μας είπε ε, επίσης αν είναι παραγωγικό ή αν είναι σκόπιμο να συζητήσουμε και το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Γιατί αν αφήσουμε αριθμίστο το θέμα και χωρίς νομοθετικές διατάξεις, αναπόφευκτα μερικές χώρες θα είναι πιο απαιτητικέ και άρα θα υποστούν τον αθέμητο ανταγωνισμό από άλλες χώρες που έχουν ε, χαμηλότερες κοινωνικές προδιαγραφές. Και κάτι άλλο που μας λέει η κυρία Μπάουρ που δεν είναι ε, η εμπνεύστη αυτής της πρότασης, αλλά επαναλαμβάνει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι το θέμα των αυτοπασχολούμενων. Τώρα, αν, ήταν, αν είχαμε θέμα αυτοπασχολούμενο και ψεύδο αυτοπασχολούμενο, θα πρέπει να είμαστε σε άλλη επιτροπή. Γιατί το θέμα αυτό συνδυάζεται άμεσα με τι οδικέ μεταφορέ. Αν εμεί συζητούμε για αυτοπασχολούμενου στη δική μα επιτροπή, είναι γιατί υπάρχουν θέματα ασφάλεια. Όχι γιατί υπάρχουν φορολογικά και οικονομικά θέματα, γιατί υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα προσωπικής ασφάλειας και ασφάλειας των πολιτών. Γιατί μιλούμε για οδηγού ε, βαρέων οχημάτων και αυτά έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια. Είπατε να μην μιλήσουμε για θέματα ανταγωνισμού μεταξύ μας. Είπατε να μιλήσουμε για αυτοαπασχολούμενου και ψευδοαυτοαπασχολούμενου. Μα δεν είναι αυτό το αντικείμενο τη Επιτροπή. Τι θα κάνουν οι σοσιαλιστέ, Οι σοσιαλιστέ θα εμείνουν στη συνένεση, στον ορθολογισμό ότι οποιαδήποτε σωματική φυσική εργασία επηρεάζει το βαθμό κόποση. Γι' αυτό και θα καταθέσουμε ουσιαστικέ τροπολογίε στην έκθεση Bauer. Και θα εμείνουμε στη συνένεση, στη συμβαστική λύση του 2002 μεταξύ Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινοβουλίου, ακόμη και νομολογίας του ΔΕΚ. Και θα μείνουμε πιστοί στην θεμελιώδη αρχή ότι όποιος και αν οδηγεί μια ταλίκα, είτε είναι αυτοαπασχολούμενος, είτε μισθωτός, είτε ψευδοαυτοαπασχολούμενος, αν είναι κουρασμένος, συνιστά κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια. Άσχετα από το ποιο είναι το νομικό καθεστώς του οδηγού. Θα δώσουμε αυτή τη μάχη μέχρι τελικής πτώσης. Και αν τα καταφέρουμε, θα κάνουμε έναν δρόμο που ήδη τον είχαμε πραγματοποιήσει το 2002. Και κρίμα που υπαναχωρήσαμε σε θέματα οδικής ασφάλειας. Αν χάσουμε αυτή τη μάχη, αν χάσουμε αυτή τη ψηφοφορία, ίσως τη χάσουμε και οριακά, τότε κυρία Μπάουερ θα αρχίσουμε να συζητούμε για αυτοαπασχολούμενος και ψεύδο αυτοαπασχολούμενος. Βέβαια θα πρέπει με το χαρακτηρισμό αυτοαπασχολούμενοι να καλύψουμε όλο τον κόσμο. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε τροπολογίες ε, είμαι είμαι εσά ή χωρί εσά, αλλά συνένεση δεν υπάρχει τώρα, κυρία Μπάουρ. Συνένεση υπήρχε το 2002. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η αρμοδιότητά μα είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και η οδική ασφάλεια των πολιτών. Εμεί, κυρία Πρόεδρε, θα εμείνουμε στη θέση μα που είναι η ιστορική θέση, κατά παράδοση θέση του Σιδερχιού, η ιστορική θέση του ΕΛΚ και η ιστορική θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φαίνεται σε όλε μα τι εκθέσει με εξαίρεση την τελευταία που λέει το ίδιο πράγμα αλλά καταλήγει σε αντίθετο συμπέρασμα. Και θα προσπαθήσουμε να το κερδίσουμε. Και αν δεν το κερδίσουμε, αν ανητηθούμε κυρία Πρόεδρε, θα υποβάλουμε ολόκληρη συστοιχεία ε, τροπολογιών, ώστε με το χαρακτηρισμό των ψευδοαυτοαπασχολούμενων να μην καλύψουμε όλους τους ε, εργαζόμενους, για να μην έχουμε και τους μισθωτούς. Γιατί τι θέλουν οι εργοδότες, για να μην υπάρχουν όρια, να τους κάνουν όλους τους ψευδοαυτοαπασχολούμενους με το ψευδοεπιχείρημα ότι έτσι θα φτάσουμε στον παράδεισο της απόλυτης και άκρατης αυτορυθ... αυτορύθμισης. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που χρειάστηκε να απουσιάσω και δεν παρακολούθησα την αρχική παρουσίαση της κυρίας Μπάουερ. Η κυρία Σρότερ και μετά η κυρία Φιγκερέντο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκφράζω εδώ την άποψη της σκιώδης ε, εισηγήτριας κυρίας Τουρούνεν. Εκείνη έχει συντάξει το έγγραφο, διότι δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα. Η σκιώδης εισηγήτριά μας, λοιπόν, αναγνωρίζει την προσπάθεια της κυρίας Μπάουερ να συντάξει μια συμβιβαστική, μια ε, γνωμοδότηση, η οποία εκφράζει την ε, συνένεση αλλά για, για μας, από τη δική μας ε, πλευρά, η συνένεση αυτή δεν αντανακλάται μέσα στο έγγραφο της κυρίας Μπάουερ δεν ε, βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο ορισμό. Αυτό το θεωρούμε σωστό, διότι αν είχε συμπεριλάβει το συγκεκριμένο ορισμό, τότε θα δυσκολουμε περισσότερα ακόμα τα πράγματα. Όμως πέραν αυτού, στο οποίο συμφωνούμε, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν μας βρίσκουν σύμφωνους συγκεκριμένα το να αφαιρέσει από, την, από το, το, σχέδιο αυτό τους αυτοαποσχολούμενους. Γιατί λοιπόν να αφαιρέσουμε αυτή την προστασία η οποία αυτή τη στιγμή προσφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί να μειώσουμε το επίπεδο της προστασίας σε συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων. Δεν καταλαβαίνω πώς θα το προωθήσουμε αυτό δεν είναι μόνο η προστασία εκείνων που οδηγούν, αλλά και όλων όσων χρησιμοποιούν τα οδικά δίκτυα, τα πεζοδρόμια, οι πεζοί, οι ποδηλάτες, οι όλοι οι πολίτες που κυκλοφορούν, όλοι αυτοί κινδυνεύουν. Αυτή λοιπόν η ε, συνολική προστασία που πρέπει να υπάρχει μειώνεται, αποδυναμώνεται. Δεν είναι αποδεκτό λοιπόν αυτό από εμά. Επίσης, οικονομικά επιχειρήματα δεν δικαιολογούν μια τέτοια μείωση. Παραδείγματο χάρη το οικονομικό επιχείρημα ενός θεμητού ανταγωνισμού. Αυτό το επιχείρημα του θεμητού ανταγωνισμού δεν καλύπτεται πλέον. Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση δεν είναι σωστή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ε, εάν κάποιος πει ότι μπορούμε να, να δεχτούμε ένα υψηλότερο ποσοστό ρίσκου όσον αφορά τα ατυχήματα και τα οικονομικά επιχειρήματα καταραίων, διότι το κόστος θα μεγαλώσει, θα αυξηθεί ασφαλώς. Όλοι λοιπόν θα χρειαστεί να επενδύσουν περισσότερο. Επίσης, μετά από αυτά που είπε ο κύριος Σέρκας, υπήρχε μεγάλο ποσοστό συνένεση σε αυτό το κοινοβούλιο ότι αυτή η οδηγία θα πρέπει να συνταχθεί έτσι, με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό κιόλας και συντάχθηκε. Πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει, είχε παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία εκπόνησης και πρέπει να πω ότι παλέψαμε σκληρά και έγιναν και πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς θα συνταχθεί η οδηγία με μία μεταβατική περίοδο, αλλά βέβαια η μεταβατική αυτή η περίοδος είχε στόχο να προσαρμοστούν και τα νέα κράτη-μέλη. Όμως όλοι είχαμε συμφωνήσει ότι κάποια μέρα θα πρέπει να παγιωθεί ένας, ε, ένα πλαίσιο θεμητού ανταγωνισμού. Και δεν νομίζω ότι αυτή η συμφωνία, αυτή η σύμπτωση απόψε, η οποία υπήρχε στο σώμα να μην υπάρχει πλέον καθόλου, να έχει εξαφανιστεί. Ε, Σας ευχαριστώ κυρία Φιγκερέντο και μετά ο κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Μας απασχολείται και πάρα πολύ καιρό. Και επίσης είναι αλήθεια ότι η μοναδική οδηγία που συγκέντρωσε ευρεία συνένεση ήταν η οδηγία του 2002, όπως ακούσαμε. Και με βάση αυτή την ευρεία συνένεση και για να καταστεί αυτή δυνατή, έγινε δεκτή μια μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή όλων των χωρών προκειμένου να συμπεριλάβουν όλες οι χώρες, όλους τους εργαζόμενους, ακόμη και τους αυτοαπασχολούμενους, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό ήταν το αντικείμενο της συνένεσης. Και μάλιστα συμμετείχα και εγώ στην συζήτηση τότε. Υπήρξε όντως ε, σημαντική συνένεση. Μερικές χώρες ζήτησαν μεταβατική περίοδο για να προσαρμοστούν στο θέμα των αυτοαπασχολούμενων. Δόθηκαν αυτέ οι μεταβατικές περίοδοι. Από το 2009 και μετά συμπεριλήφθηκαν οι πάντε, ακόμη και οι αυτοαπασχολούμενοι, στο πεδίο εφαρμογή οδηγία. Και είναι απαράδεκτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα έρχεται τώρα και να επιχειρεί αναθεώρηση και υπαναχώρηση στο θέμα αυτό. Ενώ τότε είχαμε καταλήξει συνένεση με την ε, συμφωνία τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με ε, συμφωνία και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Γιατί τώρα να ασκείται πίεση για την ε, παλινδρόμηση. Και ορισμένοι βουλευτές του ΕΛΚ, αλλά όχι μόνο του ΕΛΚ, θέλουν να καλύψουν ορισμένες οργανώσεις μεταφορών που θέλουν να, να διατηρήσουν μια ανυπόφορη κατάσταση και δίνουν πρωταρχική σημασία στο κέρδος τους εις βάρος όλων των υπόλοιπων παραγόντων, εις βάρος των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμορφώνονται με την οδηγία, εις βάρος της ασφάλειας και των οδηγών, των εργαζομένων και των υπόλοιπων επιβατών, εις βάρος της υγείας των οδηγών, αλλά πάνω απ' όλα εις βάρος της ίδιας της οδικής ασφάλειας. Γιατί το, το ξέρουμε όλοι, ότι όταν είμαστε κουρασμένοι, οδηγούμε μηχανικά. Δεν έχουμε τη δέουσα επαγρύπνηση και προσοχή. Είναι φυσιολογικό όταν κάποιος είναι κουρασμένος να μην έχει όλες τις αισθήσεις εγρήγορση. Η κυρία Μπάουερ έγινε φερέφων αυτών των θέσεων που είναι γνωστές, ήταν γνωστές από παλιά, αλλά μετά από εκτενείς συζητήσεις ε, σιώπησαν. Τώρα ξαναβήκα στην επιφάνεια όλες αυτές οι απόψεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις περιπτώσεις κοινωνικού dumping. Ας μην ξεχνούμε ότι δεν μιλούμε εδώ για ψευδό μόνο υπό φορολογική άποψη, υπό το φορολογικό πρίσμα. Μιλάμε για θέματα δικής ασφάλειας πάνω απ' όλα και υγείας των εργαζομένων. Για να διατηρήσουμε την ισορροπία του κειμένου, θα πρέπει να εμείνουμε στην αρχική οδηγία του 2002, αμετάβλητη, και να συμπεριλάβουμε και τους αυτοαπασχολούμενους από πέρυσι στο πεδίο εφαρμογή οδηγία. Γιατί τώρα να απορριθμίσουμε αυτό που ήδη είχαμε ρυθμίσει. Δεν έχω άλλο επιχείρημα, δεν χρειάζεται να, να προσθέσω τίποτα άλλο γιατί οι συνάδελφοι Σέρκας και Σρέντερ παρουσίασαν πολλά επιχειρήματα, αρκετά εμπεριστατωμένα. Νομίζω το θέμα είναι φως φανάρι. Έχουμε και την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Πάντως για μένα το πρωταρχικό ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε αμετάβλητη την αρχική οδηγία που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους και θα συμπεριλαμβάνει στο πεδίο της και τους αυτοαπασχολούμενους. Ο κύριος Τόμας Μάν μετά η κυρία Μαριάν Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Edith Bauer προσπάθησε πράγματι να βασίσει την ε, έκθεσή της σε μια συνένεση, σε, μια, σε συνενετικές απόψεις. Όμως ε, είναι αδύνατον, και εδώ βλέπουμε ε, σε περιορισμένο χρόνο, να επιτύχουμε μία σύμπτωση απόψεων μεταξύ μας. Η κυρία ε, Φιγκουερέιδο είπε ότι και στο παρελθόν Έχουμε ασχοληθεί με αυτό το καυτό θέμα και η κυρία Σρούντερ το είπε, αλλά εν τέλει ασκήσαμε χρονική πίεση στην εισηγήτρια και κάναμε, την κάναμε ταχογράφο. Δηλαδή της είπαμε, προχώραμε με μια μεγάλη ταχύτητα ε, και ενώ το θέμα μας, το σοβαρό αυτό θέμα είναι να έχουμε συγκεκριμένο χρόνο ε, εργασίας ε, των οδηγών ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνθήκων εργασίας ε, που να αποφεύγει το, τους κινδύνους σε περίπτωση που είναι κουρασμένοι κλπ. Ε, βεβαίως οι επιχειρήσεις είναι ανταγωνιστικές. Εξέτασα τρεις επιχειρήσεις τέτοιες οδικών μεταφορών, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μια μικρομεσαία και ένα, μία επιχείρηση την οποία επισκέφθηκα μία φορά και δεν θα ξαναεπισκεφθώ ποτέ διότι τα πάντα μέσα σε αυτή την συγκεκριμένη εταιρεία ήταν στραβά. Λοιπόν, έρχονται παραγγελίες, ε, γίνονται προσπάθειες να υπονομεύσει ο ένας ανταγωνιστής τον άλλον και στη συγκεκριμένη κακή εταιρεία, την τρίτη δηλαδή που σας είπα, ε, είχα την εντύπωση ότι υπήρχε φοβερή πίεση πάνω στους οδηγούς να δουλέψουν περισσότερο, να οδηγήσουν περισσότερες ώρες και αν, δηλαδή εκβιαστικά τους πίεζαν και αν δεν συμμορφώνονταν τους πετούσαν έξω από την εταιρεία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ε, να ε, επιτύχουμε, να, να, να, να, ρυθμίσουμε τα πάντα όταν υπάρχουν τέτοιες διαφορές στην αγορά εργασίας των εταιριών αυτών. Βεβαίως έχω δει και πάρα πολλές εταιρείες που λειτουργούν ικανοποιητικά και μερικές εξαιρετικά καλά. Ε, οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε, σε αυτές τις ε, οδικές μεταφορές δεν είναι μόνο κίνδυνοι για τους οδηγούς ή τους επιχειρηματίες, είναι κίνδυνοι για όλους μας. Η κυρία Μπάουερ νομίζω ότι πολύ σωστά ανέφερε ε, την τροπολογία 12. Μην ξεχνάτε ότι η Κομισιόν ήθελε να το εδάφιο 12. Μην ξεχνάτε ότι η Κομισιόν ήθελε να διαγράψει το ε Λοιπόν, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μία ε, ε, σαφήνεια στους ορισμούς και καλώς συμπεριέλαβε τους αυτοαποσχολούμενους. Έχω ε, πρόβλημα με την τροπολογία 6, η οποία αναφέρει κάτω από 3,5 τόνους. Δηλαδή είναι τα μικρά φορτηγάκια που χρησιμοποιούν εταιρείε διανομής πίτσας, μικρά φορτηγά. Ε, χρήσεως βάρους κατωτέρου των 3,5 τόνων. Πώς μπορούμε να το δικαιολογήσουμε αυτό. Εδώ έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ίσως μπορέσει να μου απαντήσει η κυρία Μπάουερ. Και η τροπολογία 13. Επίσης μου δημιουργεί πρόβλημα. Εδώ έλεγε ότι δεν θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι που δημιουργούν διακρίσεις. Τι εννοεί αυτό, μη, διακριτικές, ε, μη διακριτική έλεγχη, τι εννοεί. Δεν θα ελέγξουμε όλες τις χώρες, θα ελέγξουμε μόνο ορισμένες χώρες ή θα εξαιρέσουμε ορισμένους κλάδους ε, για να μην γίνουν διακρίσεις. Αυτό πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Θα ήθελα λοιπόν να μου το διευκρινίσει αυτό, τι σημαίνει η επιβολή ελέγχων που δεν δημιουργούν διακρίσεις, non-discriminatory, ε, για να μπορέσουμε με, ησυχή, με ασφάλεια να ελέγξουμε και να υποπτεύσουμε το τομέα αυτό των οδικών μεταφρών, αλλά και να κυκλοφορούμε στους δρόμους με το αίσθημα της ασφάλειας. κυρία Μαριάννα και μετά ο κύριος Κομφεράτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμβιβαστικό κείμενο και νομίζω ότι η κυρία Μπάουρ έχει κάνει μία προσπάθεια. Παρακολούθησα με προσοχή τη συζήτηση και αναρωτιέμαι εάν ένας συμβασμός είναι δυνατό να γίνει. Θα επανέλθω όμως. Εδώ ο στόχος μας είναι να αναθεωρήσουμε την οδηγία 2002 και να συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι. Ξέρω ότι πολλά, πολλοί συνάδελφοι ρώτησαν γιατί θέλουμε να την αλλάξουμε. Γεγονός είναι ότι τα πράγματα εξελίσσονται, έχει και η Κομισιόν αλλάξει πολλές φορές την άποψή, τους, την άποψή της. Εάν εμείς λοιπόν οι νομοθέτες δεν λάβουμε υπόψη τις αλλαγές που έχουν γίνει, δεν εκτελούμε σωστά το έργο μας. Άρα λοιπόν υπάρχει νόμιμη δικαιολογία, νόμιμος λόγος για τον οποίο θέλουμε να κάνουμε την αναθεώρηση. Κανένας όμως δεν μου έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι ειδικά οι αυτοαπασχολούμενοι είναι πιο επικίνδυνη από τους ε, μισθωτούς απασχολούμενους, ε, από τους μόνιμους, από τους ε, απασχολούμενους σε εταιρείες, υπαλλήλους. Δεν έχω λοιπόν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Όταν τα στοιχεία για τα ατυχήματα δεν διακρίνουν μεταξύ αυτοαπασχολούμενων και μη αυτοαπασχολούμενων και πιστεύω ότι αυτό είναι ακριβώς και το σημείο της αντιπαράθεσης για την συμπερίληψη ή όχι των αυτοαπασχολούμενων. Επίσης, η η κούραση είναι ένας παράγων, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει ομοίως να συμπεριληφθούν. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Σέρκας και είπε ότι θα πρέπει όλος ο χρόνος, όλη η εργασία να ληφθεί υπόψη σαν μετρήσιμο στοιχείο. Τότε, αν το υιοθετήσουμε αυτό σημαίνει ότι κάθε οδηγός ο οποίος απασχολείται, είναι υπάλληλο δηλαδή, δεν θα μπορέσει να εκτελεί καμία μερική εργασία πουθενά αλλού. Παραδείγματο χάρη, δεν μπορεί να πάει στο καφενείο του αδελφού του και να σερβίρει καφέδες. λοιπόν κάθε επιπλέον πλέον η διαφορετική εργασία πλην της σταθερής του απασχόλησης. Ακούω ήδη πολλούς ε, ψιθύρους και επιφυλάξεις. Αλλά υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εάν συμπεριλάβουμε τους αυτοαποσχολούμενους οδηγούς, η πραγματικότητα σημαίνει ότι εάν κάποιος ε, φύγει από το, ε, το πάρκινγκ της εταιρείας, αφήσει το φορτηγό του και πάει στο σπίτι του, και εν συνεχεία πάει, όπως είπαμε, στο καφενείο του αδελφού του, πώς θα τον ελέγξουμε. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να τον ελέγξουμε είναι τον, αν τον αστυνομεύσουμε από τη στιγμή που κλείνει την πόρτα του φορτηγού του, πηγαίνει στο σπίτι του και να δούμε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί τι κάνει. Υπάρχουν λοιπόν δυσκολίες, παρακολούθηση δυσκολίες ελέγχου. Επίσης υπάρχουν και στοιχεία υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Δεν έχω δει λοιπόν από πουθενά εμ, πραγματικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι οι αυτοαπασχολούμενοι είναι πιο επικίνδυνοι από τους ε, άλλους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας. Πιστεύω λοιπόν ότι ακόμα και αν συμπεριλάβουμε τους αυτοαπασχολούμενους και δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας αυτής της εργασίας, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτύχουμε ένα συμβιβασμό, ένα συγκερασμό απόψεων. Αυτοί, και κάτι άλλο, αυτοί που πραγματικά αυτοαποσχολούνται, που είναι σωστοί επιχειρηματίες, θα τους ε, ζημιώσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Θα βλαφτούν διότι τους μεταχειριζόμαστε σαν παιδιά και εμείς ε, είμαστε ας πούμε σαν ταντάδες των παιδιών αυτών και δεν τους αφήνουμε καμία πρωτοβουλία και ευελιξία. Ο κύριος Κομφεράτη. Ευχαριστώ. Ακούσα για μία ακόμα φορά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα μας είπε η κυρία Μπάουερ. Όμως, ειλικρινά, στην ε, έκθεσή της ε, δεν βλέπω κανένα πλαίσιο αναφοράς που να επιτρέπει επίτευξη ε, συμφωνία, συμβιβαστική συμφωνία. Το αντίθετο μάλιστα. Εάν πρέπει να κάνουμε οδηγία, θα πρέπει να καθορίσουμε πρώτα ποια προβλήματα θα πρέπει να λύσει αυτή η οδηγία, τι στόχους θα πρέπει να έχει. Εγώ πιστεύω ότι τα προβλήματα προς επίλυση είναι δύο. Το πρώτο αφορά την ασφάλεια υπό το φως των δεδομένων και των στοιχείων τα οποία έχουμε και υπό το φως των θεωρήσεων και των σκέψεων που ακούσαμε εδώ από τους ενδιαφερόμενους ε, που αυτό απασχολούνται ή είναι υπάλληλοι στον κλάδο αυτό. Γιατί ε, ε, εδώ μιλάμε μόνο για την ασφάλεια των πολιτών που μπορεί να ε, έχουν πρόβλημα να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εδώ παίζεται και η ασφάλεια των εργαζομένων, γιατί αν ε, ο εργαζόμενος δεν δουλεύει με καλές συνθήκες, τότε κινδυνεύει να χάσει την ίδια του τη ζωή ποιες είναι οι βέλτιστες ε, συνθήκες, έτσι ώστε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες να κάνει κανείς τη δουλειά αυτή. Ποια είναι τα εργαλεία της δουλειάς. Είναι πρώτα απ' όλα τα οχήματα, άρα τεχνολογικά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες εργασίας αντικειμενικά να είναι σωστές. Πιστεύω λοιπόν ότι το πραγματικό πρόβλημα ε, ξεκινάει από, τους αρνητικ... από τις αρνητικές συνθήκες στις οποίες καλείται ο εργαζόμενος να εργαστεί. Και εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Ένα ζήτημα είναι ο χρόνος εργασίας η ποσότητα των ωρών ε, που εργάζεται ο εργαζόμενος. Αυτό ισχύει για όλους τους εργαζόμενους και για μας ακόμη. Επομένως, όσο περισσότερες ώρες εργασίας και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να το καταλάβει κανείς ακόμα και αν δεν είναι γιατρός και εν πάση περιπτώσει ο κάθε γιατρός θα σας το εξηγήσει ότι κάθε ώρα επιπλέον εργασίας που προστίθεται τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο οδηγός, ο εργαζόμενος. Δεύτερον, η ένταση της εργασίας. Ε, υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να μην ε, διαρκούν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά όμως είναι ιδιαίτερως κουραστικές γιατί απαιτούν μεγάλη συγκέντρωση και επομένως ξεπέρασμα κάποιων ωρών εργασίας μπορεί να σημαίνει μείωση αντανακλαστικών κλπ. Σας δίνω πολύ απλουστευτικά παραδείγματα, αλλά αυτό που είναι ότι η ασφάλεια μπορεί να έχει πολλά ε, στοιχεία συνθετικά, όμως όλα τα στοιχεία αυτά τα βρίσκουμε στους μετακινούμενους εργαζόμενους. Επομένως, ασφάλεια του οχήματος, ε, καλές συνθήκες εργασίας, ένταση και ε, ε, μεγάλο διάστημα οδήγησης. Ας πούμε, εάν είσαστε σε ένα όχημα το οποίο ε, του οποίου τα παράθυρα κλείνουν και κλείνουν καλά, ε, τότε δεν θα έχετε πρόβλημα. Εάν βρίσκεστε σε ένα όχημα του οποίου τα παράθυρα μένουν ανοιχτά για κάποιο λόγο, τότε πολύ γρήγορα θα έχετε ένα αίσθημα κόπωσης. Επίσης, ασφάλεια όλων αυτών που οδηγούν σε ένα διπλανό όχημα, το οποίο, με το οποίο μπορεί να ε, συγκρουστεί το εν λόγω όχημα του εργαζόμενου. Ε, υπάρχουν ε, οι, αυτοί που περπατούν ε, δίπλα στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο κτλ. Όμως, έχουμε και τους ίδιους τους εργαζόμενους που εργάζονται σε κάποιες επιχειρήσεις. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα του κοινωνικού dumping. Και ε, μιλάμε εδώ για απασχόληση η, της οποίας ε, ο μισθός ε, δεν εξαρτάται από το πόσο καλά κάνεις τη δουλειά σου, αλλά από το γεγονός ότι τη δουλειά που κάνεις εσύ είναι διαθέσιμη πάρα πολύ να την κάνουν. Επίσης, αυτοί οι πολλοί είναι διατεθειμένοι να την κάνουν με πολύ διαφορετικές συνθήκες από ό,τι την κάνεις εσύ. Και επομένως εγώ λέγω ότι θα πρέπει να υπολογιστούν και οι αυτοαπασχολούμενοι αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι εταιρείε του κλάδου ε, θα πρέπει να ε, μας απασχολήσουν. Και εν πάση περιπτώσει δεν λύνουν τα πράγματα εάν κάνουμε, αν γράψουμε ε, μία οδηγία ή δύο. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο όρος ψευδοαυτοαπασχολούμενος έχει εφευρεθεί έτσι ώστε να βρεθούν παραθυράκια στον νόμο. Εάν όλοι έχουν ε, απέναντί τους τις ίδιες προϋποθέσεις, τις ίδιες απαιτήσεις και τις ίδιες συνθήκες, τότε δεν χρειάζεται να δεν θα υπάρχει λόγος να προστρέξει κανείς σε αυτό το ψεύτικο επιχείρημα του ψευδοαυτοαπασχολούμενου. Γιατί διαφορετικά πάντα στου εργαζόμενου στους εργαζόμενους αυτούς και σε αυτόν τον τύπο εργασίας θα υπάρχουν πάντα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαυνόρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πάουερ για την ε, εργασία της, ε, πολύ σκληρή εργασία για να προετοιμάσει την έκθεση. Να την ευχαριστήσω για το θάρρος ε, και την εντιμότητά της. Γνωρίζουμε όλοι ότι η συνένεση σε αυτόν τον κλάδο είναι δύσκολη, βλέπε αδύνατη. Το παράδειγμα έχει δοθεί ήδη από την οδηγία για τον χρόνο εργασίας, επί της οποίας δεν εξευρέθη συνενετική λύση. Συμφωνώ, στηρίζω την κυρία Μπάουερ όταν λέει ότι το να βρούμε μια λύση είναι πιο σημαντικό από το να έχουμε οπωσδήποτε συμβιβαστική λύση και λέω ότι ενδεχομένως θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία και άρα λύση. Πολλές επικρίσεις ακούστηκαν όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας. Πιστεύω ότι οι σόφρονες γνωρίζουν και αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Η Κομισιόν αναγνώρισε το λάθος της και προσπάθησε να επιφέρει διορθώσεις. Και γι' αυτό λοιπόν μας υποβάλλει το ε, το σχέδιο το οποίο έχουμε σήμερα ενώπιόν μας. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το σύνολο της οδηγίας. Ήδη κάποιος συνάδελφος είπε ότι πρέπει να σκεφτούμε τον λόγο ύπαρξης αυτής της οδηγίας, γιατί υπάρχουν δύο θέματα τα οποία αναμειγνύονται στην οδηγία αυτή. Το ένα είναι ο χρόνος εργασίας των εργαζομένων και το άλλο θέμα είναι η οδική ασφάλεια. Πρόκειται λοιπόν για δύο θέματα τα οποία δεν συνδέονται απαραίτητος, έστω και αν και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Όσον αφορά το θέμα των αυτοαπασχολούμενων και των ψεύδο αυτοαπασχολούμενων, θέμα πάρα πολύ σημαντικό φυσικά, δεν περιορίζεται στον τομέα των οδικών μεταφορών. Το πρόβλημα των ψεύδο ή πραγματικών αυτοαπασχολούμενων αφορά ένα σωρό κατηγορίες εργαζομένων, όχι μονάχα τους οδηγούς, αλλά ε, και ένα σωρό άλλους εργαζόμενους, νοσοκόμους κτλ. Όσον αφορά τώρα τη διαμόρφωση του χρόνου εργασίας και αυτός και αυτό το θέμα δεν συνδέεται με το, τις οδικές μεταφορές. Όταν απειλείται η ζωή σου από ένα όχημα, δεν σε ενδιαφέρει αν το όχημα αυτό το οδηγεί ένας αυτοαπασχολούμενος, ένας ψευδοαπασχολούμενος ή ένας οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος. Και ξέρουμε ότι οποιοδήποτε ε, οδηγήσει πολλές ώρες, ε, ε, φυσικά δεν θα μπορεί να οδηγήσει αλλά ξέρετε, κατά αυτήν την έννοια θα έπρεπε να πούμε σε κάθε Ευρωπαίο εργαζόμενο, αν έχεις δουλέψει 8 ή 9 ώρες στο γραφείο σου, δεν μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητό σου για να γυρίσεις στο σπίτι σου, γιατί είσαι επικίνδυνος οδηγός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή τη ρητορική σας δυνότητα. Η κυρία Γκρινή και μετά ο κύριος Χάντελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα παρόλα αυτά να συγχαρώ την Edith Power γιατί χρειάζεται μεγάλο κουράγιο και τόλμη για να πραγματευτεί κανείς αυτό το θέμα. Αυτά εισαγωγικά, αν και οι παρατηρήσεις μου δεν θα είναι εξίσου εγκομιστικές και για το κείμενο. Είναι δύσκολο αυτό το θέμα για τους αυτοαπασχολούμενους, γιατί εξορισμού ε, ισχύει η ελευθερία εργασίας και ο περιορισμός των αυτοαπασχολούμενων είναι δύσκολο πράγμα. Φυσικά, έχουμε υπόψη τη οδική ασφάλεια, είναι δική μας αρμοδιότητα και να σκεφτούμε και τον αθέμητο ανταγωνισμό. Ε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων. Όταν μου λέτε ότι είναι δύσκολο να υπολογίσουμε το χρόνο εργασίας τους, μπορούμε να εργαστούμε με κάποιους ελάχιστους χρόνους. Να υπολογίσουμε το χρόνο οδήγησης, αυτό γίνεται εύκολα, το χρόνο φόρτωση εκφόρτωσης και για το διοικητικό σκέλος, που είναι όντως δύσκολο να αξιολογηθεί, θα μπορούσαμε να, προσ... να προσθέσουμε ένα καταποκοπή χρόνο και έτσι να καταλήξουμε σε ένα ελάχιστο χρόνο εργασίας που πραγματοποιήθηκε. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο αυτό. Διάβασα με προσοχή τις τροπολογίες και αντιλαμβάνομαι ότι για να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις η τροπολογία 5 που λέει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής οδηγίας Έχουμε πει όμως ότι αυτή η ε, διάδεξη δεν θα παραβλέπει το δικαίωμα των κρατών μελών ε, να υποβάλουν κάποιες νομοθετικές διατάξεις. Να πούμε δηλαδή εμείς στη Γαλλία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να μας δώσουν το χρόνο εργασίας τους, ενώ πώς θα ελέγξουμε τους Βέλγους για παράδειγμα. Είναι δύσκολο. Αν αποκλείσουμε τους ψεύδο αυτοαπασχολούμενους, πώς θα ελέγξουμε την κατάσταση. Ένας οδηγός διασχίζει ολόκληρη τη Γαλλία θα το σταματήσουμε και πώς θα υπολογίσουμε το χρόνο εργασίας του για να τον χαρακτηρίσουμε ψεύδο αυτό που ασχολούμαι. Αυτό είναι αδύνατο. Λυπούμε, λυπούμε, αλλά δεν συμφωνώ με την έκθεση της κυρίας Μπάουερ. Και πολύ λυπούμε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσάμπρνοχ ζήτησε το λόγο για διαδικαστικό. Πολύ ευχαριστώ. Σας ακούμε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπερασπίσω τον εαυτό μου απέναντι στο σχόλιο σας, το ηρωνικό για τη ρητορική μου δυνότητα. Ε, εγώ είχα εκτενείς διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Μεταφορών, με κοινωνικούς εταίρους. Σας θέρμα παρακαλώ λοιπόν να αποφύγετε τέτοιου είδους προσωπικούς επενιγμούς. Mm. σημειώνω το διαδικαστικό. Εντάξει, προσπαθώ να προεδρεύσω αμερόληπτα Μερικές φορές όμως δεν μπορώ να κρατηθώ. Είμαι κι εγώ πολιτικός και αντιδρώ ενθερμό. Αυτή βέβαια είναι η προσωπική μου γνώμη. Δεν έκανα το σχόλιο ως πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και δικαίως το επισημαίνεται, κύριε Κάμπρνοχ. Το λόγο έχει ο κύριος Χέντελ και μετά ο κύριος Σόρι. Κύριε Σέρκας, και εσείς διαδικαστικό θέλετε. Εκτό μικροφόρου δυστυχώ, στο σχόλιο του κ. Σέρκα. Καλώ θα σα δώσουμε το λόγο, αλλά στο τέλο, γιατί ήδη έχετε μιλήσει, και εκεί πραγματικά θα είμαι αδιάλεκτη. Ο κ. Χέντελ. και αν σα δώσω το λόγο τώρα, τότε είναι που θα με κρίνουν υποκειμενική και μεροληπτική πρόεδρο και αυτό θα είναι πραγματικά αντιπαραγωγικό για την Επιτροπή μας. Ο κ. Χέντελ και μετά ο κ. Σόρη. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι υποστηρίζω τη συνάδελφό μου, κυρία Φιγκουερέντο, αλλά και η κυρία Σρέντερ και ο κύριος Σέρκας. Θα ήθελα να φερθώ σε δύο πτυχές. Πρώτο σχόλιο αφορά τον κύριο Μαν και συνεχεία τη συνάδελφο κυρία Χάρκιν. Σε... Όσον αφορά αυτή την έκθεση Bauer πρέπει να εκτιμήσουμε δύο στοιχεία. Πρώτον ότι έγινε μια πραγματική προσπάθεια ορισμού του τι είναι αυτοαπασχολούμενος ε, και τι είναι ε, μία αυτοαπασχολούμενος. Πώς θα πρέπει λοιπόν ένας ε, ε, ικανός αστυνομικός ή μάλλον τροχαίος να αξιολογήσει την, ε, και να εφαρμόσει τους κανονισμούς στο δρόμο όταν, κάνουμε, όταν δεν έχουμε σαφείς ορισμούς. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν το καθήκον να συντάσσουν δίκαιους νόμους και εάν δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει δίκαιη νομοθεσία πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς να επιβάλλουμε καλύτερους και περισσότερους ε, τροχαίους και οδικούς ελέγχους, όχι λιγότερους. Τώρα ε, απευθύνουμε στον κύριο Μαν. Έχει διαφορά εάν κάποιος είναι ανταγωνιστικός ή αν κάποιος υπονομεύει, υποσκάπτει τους ανταγωνιστές τους. Εάν κάποιος ενεργεί βρώμικα, τότε μπορεί να κατηγορηθεί ποινικά, θα πρέπει να ειδοποιηθεί η αστυνομία κλπ. Έχει λοιπόν ουσιαστική σημασία εάν ο νομοθέτης καλύπτει τον αθέμητο ανταγωνισμό ή δεν τον καλύπτει. Διότι άλλο θεμητός ανταγωνισμός, άλλο αθέμητος ή βρωμικο ανταγωνισμός. Θα έχει λοιπόν ουσιαστική σημασία αν καλύπτεται και, και ο αθέμητος ανταγωνισμός από τον νομοθέτη για την προστασία του σωστού ανταγωνισμού. Τρίτον, προς τον κύριο Μάν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι διατάξεις τις οποίες υιοθετήσαμε εμείς στο Κοινοβούλιο έχουν πλέον ακυρωθεί διότι έχουν βγει καινούργια οχήματα κάτω από 3,5 τόνους. Είναι λοιπόν κενές περιεχομένου πλέον αυτές οι διατάξεις. Εάν αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπω μικρά φορτηγά τα οποία τρέχουν ηλικιωδώς με 190 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, πραγματικά ταράζομαι ιδιαίτερα τρέμω και φοβάμαι. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε λογικά μέτρα ελέγχου σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουν γίνει στους δρόμους. Ε, πολλά άλλα πράγματα έχουν αλλάξει από το παρελθόν στο παρόν. Γνωρίζουμε περισσότερα επιστημονικά στοιχεία ε, γνωρίζουμε περισσότερα για την, τους απασχολούμενους, για την αγορά εργασίας, γνωρίζουμε για το χρόνο εργασία τους και όλες αυτέ, όλη αυτή μας η προσπάθεια δεν αφορά μόνο τους οδηγούς αλλά και το περιβάλλον και όλους αυτούς που θίγονται από τα ασφάλματα οδηγών οι οποίοι δημιουργούν ατυχήματα επειδή έχουν δουλέψει υπερβολικές ώρες. Αφορά και όλους τους θυγόμενους. Υπάρχει λοιπόν διαφορά Εάν ένας ευρωβουλευτής εδώ το κοινοβούλιο ε, λέει διάφορες ανοησίες στο τέλος της ημέρας επειδή είναι κουρασμένος, αλλά εάν ένας φορτηγατζής την τελευταία ώρα της δουλειάς του που είναι πτώμα, δημιουργεί, είναι υπέτειος ενός ατυχήματος, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οι ευθύνε είναι πολύ μεγαλύτερες. Φοβούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε σήμερα στο τραπέζι μας καλύπτει ένα μικρό μέρος του όλου προβλήματος. και ακολουθεί τη γραμμή της Κομισιόν. Δηλαδή, να μειώνει την ουσία ε, της ρύθμισης των ορών εργασίας ως συστατικό της πολιτικής ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Αυτή την πολιτική ακολούθησε η Κομισιόν εδώ και χρόνια. Εδώ προσπαθούμε να εδραιώσουμε ένα δίκτυο ασφάλειας, προστασίας. Αυτό θέλουμε να επιβάλλουμε και πιστεύω ότι θα πρέπει να όλοι να προβάλλουμε λογικά επιχειρήματα. Ο Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικής φύσεως παρατηρήσεις. είναι γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τους ψευδοαυτοαπασχολούμενους και τους πραγματικούς αυτοαπασχολούμενους. Καλά, κατά την άποψή μου, αυτό το δίλημα είναι ε, ψευδές. Ε, δεν μας ενδιαφέρει τι καθεστώς έχει ο κάθε οδηγός, μας ενδιαφέρει τι είδους εργασία κάνει και νομίζω ότι ακόμα και εδώ μέσα στο κοινοβούλιο μπορώ να σας δείξω ένα σωρό ψεύδο αυτοαπασχολούμενους. Επομένως δεν μας ενδιαφέρει το καθεστώς των εργαζομένων, αλλά μας ενδιαφέρει το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, το πώς δουλεύουν. Ξέρουμε ότι μερικές φορές ε, κάποιος εργαζόμενος ε, αποφασίζει να γίνει αυτό που λέμε ψεύδο αυτοαποσχολούμενος έτσι ώστε ε, να επωφεληθεί από κάποιες διατάξεις, συνθήκες κτλ. Θα ήθελα να ασχοληθούμε να ασχοληθώ επίσης με το προηγούμενο. Σε ένα τομέα όπου υπάρχουν ισχύουσες διατάξεις για προστασία, για ασφάλεια, υπάρχουν ταχογράφοι, υπάρχουν ε, συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένοι κανόνες όσον αφορά τους, ε, το χρόνο εργασία, τις ώρες οδήγησης, τις ώρες ξεκούρασης κτλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση για αυτές τις λεπτομέρειες που αναφέρονται εδώ ε, και σχετικά με το εάν θα πρέπει τους αυτοάποσχολουμένους να τους θεωρήσουμε μισθωτούς. Τρίτον, πιστεύω ότι δεν πρέπει επίσης να ε, υπερνομοθετούμε γιατί όταν ε, έχουμε τόσο ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο ή μάλλον όταν υπερνομοθετούμε καμιά φορά δεν καταλαβαίνουν και οι πολίτες της Ευρώπης τι ακριβώς ε, κάνουμε και δεν καταλαβαίνουν ε, ε, τι γίνεται με την έννοια ότι μετά τα κράτη-μέλη δεν πρόκειται να σεβαστούν τους νόμους αυτούς και τους κανονισμούς αυτούς. Ε, και πολύ συχνά, ξέρετε, υπερνομοθετώντας, θεσπίζουμε ε, κανόνες οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν είναι εφικτοί, δεν, είναι, ε, δεν εφαρμόζονται. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και να διατηρηθεί η νομική ασφάλεια γιατί διαφορετικά ε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σωστή διαχείριση του δικού μας χρόνου εργασία. Θα, κάνω ένα σχόλιο. Ευτυχώς απουσιάζει ο κύριος ε, ε, Καβρνόχ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρή. Και τελείως μεροληπτικά θα δώσω το λόγο στον κύριο Σέρκας, γιατί θα είναι σύντομος. Η κυρία Μογά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν και εγώ θα ήθελα να επενέσω, όπως έκανε και η κυρία Πασκάλ Μπρινή στην φίλη μας Edith Power, γιατί πραγματικά είχε το κουράγιο και την τόλμη να επομιστεί αυτή την έκθεση που είναι πολύ άχαρη. Και δεν υπήρχαν και πολλοί επίδοξοι μνηστήρες για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να την ευχαριστήσω ειλικρινά, γιατί δεν είναι καθόλου ασήμαντο αυτό το θέμα. Και εύκολο. Κάποιος ε, υπενήχθηκε ότι στο ΕΛΚ υπήρξαν απαράδεκτες πιέσεις. Θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με τη θέση της Edit Power, αλλά σε καμία περίπτωση που δεν είχαμε πιέσεις ε, προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Και στο ΕΛΚ όλοι μας έχουμε ελευθερία έκφρασης των απόψεων όμω μερικέ μερικές φορές είναι και διστάμενος. Όσοι πενήσονται ότι στο ΕΛΚ ασκούνται ανυπόφορε πιέσεις, το διαψεύδω ριζικά. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του και την ελευθερία έκφρασης. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να επιμείνω σε ένα θέμα Κατάγομαι από μια περιοχή που μονίμως βλέπει ατέλειωτες πομπές ε, τριαξονικών να διασχίζουν την Ευρώπη και να διανύουν τεράστιες αποστάσεις. Και δυστυχώς είχαμε πολύ σοβαρά τροχέα στους αυτοκινητοδρόμους μας ε, που είχαν πολύ σημαντικό αντίκτυπο Γι' αυτό και ο κόσμος είναι πολύ ευαίσθητος ε, για τις πολιτικές μας επιλογές στο θέμα των οδικών μεταφορών. Και οι πολίτες μας ενθαρρύνουν να λάβουμε πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια. Και ας μην ξεχνούμε ότι τη στιγμή που συζητούμε αυτή την έκθεση έχουμε και προσπαθούμε να, προσα... να προαγάγουμε εθνικές συντονισμένες πολιτικές για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για τους ε, οδηγούς των μεταφορών. Δεν θυμάμαι ποιος είπε πριν, αλλά και οι ιδιώτες ε, έχουν ατυχήματα μερικές φορές όταν είναι κουρασμένοι, όταν έχουν εργαστεί. Όντως. Αλλά όταν επιστρέφει κανείς ε, στο σπίτι του ε, όσο κοντά και αν είναι, τότε είναι που έχουμε την αιχμή των ατυχημάτων. Είναι πραγματικό θέμα λοιπόν οδικής ασφάλειας. Οι οδικές μεταφορές ε, μεγάλων αποστάσεων δεν μπορεί να ξεφύγει από τον κανόνα αυτό. Και όταν μάλιστα ε, οδηγεί πολύ συχνά σε αυτοκινητοδρόμους με φορτηγά και τριαξονικά και βλέπει οδηγούς να ασχολούνται και με άλλα θέματα με άλλα πράγματα και μάλιστα ε, επικαλούμε εδώ ένα άρθρο σε εφημερίδα ε, έγινε αλλαγή οδηγού σε ε, όχημα εν κινήσει που έτρεχε με 130 χιλιόμετρα την ώρα και αυτό ε, το ανακάλυψε ένας αστυνομικός την ώρα που έτρεχε δίπλα στο το τριαξονικό γινόταν αλλαγή οδηγού από τον ένα στον άλλον, ενώ το όχημα δεν σταμάτησε καν. Αυτό είναι πραγματικά μείζον θέμα δική ασφάλεια. Ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι όλοι προσπαθούμε να χτίσουμε από κοινού την κοινωνική Ευρώπη. Και η παλινδρόμηση σε σχέση με μία διάταξη του 2002 που ίσχυε μέχρι το Μάρτιο του 2009 μοιάζει με υπαναχώρηση σε σχέση με τα κεκτημένα της κοινωνικής Ευρώπης. Είναι σαν να ακυρώνουμε ένα σημαντικό έργο που επιτελέσαμε στην Επιτροπή μας και να το ματαιώνουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο χρόνος εργασίας ήταν ένα σημαντικό θέμα συζήτησης. Ο χρόνος εργασίας, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στους θέσεις εργασίας τους, η καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, Όλα αυτές οι αρχές και όλα αυτοί οι στόχοι μας καθοδηγούν. Είναι η πολιτική μας πηξίδα. Υπάρχει και, και το πολιτικό και το οικονομικό βέβαια ζήτημα. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε κάποιες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή να υποστηρίξουμε κάποιες διατάξεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενθαρρύνουν τον αθέμητο ανταγωνισμό και που μάλιστα ε, είναι και επίμαχες. Και αυτό από σεβασμό προς τον επαγγελματικό κλάδο των μεταφορέων και από σεβασμό προς τα συνδικάτα που συναντήσαμε στην ομάδα εργασίας που προεδρεύουμε τον Αλεχάνδρο, γιατί είχαμε διαβουλεύσει με εκπροσώπους συνδικάτων για το θέμα αυτό. Εγώ λοιπόν διαφωνώ με την έκθεση αυτή, γιατί περιλαμβάνει κάποια σημεία που δεν είναι συνενετικά. Και για έλεγχο, μην μου μιλάτε εμένα για έλεγχο. Ανήκω σε ένα επαγγελματικό σώμα ελέγχου και είναι πολύ δύσκολος ο έλεγχος, γιατί όπως είπε η Πασκά Γκρενιά, ακόμη πιο δύσκολος είναι σε τέτοιου είδους εργαζόμενους. Και μιλήσαμε για τα φορτικά κάτω των 3,5 τόνων, μη μιλήσατε για τους ε, πιτσαδόρου. Ε, ή τους οδηγούς τροχόσπιτων και αυτοί εμπίπτουν. Είναι οχήματα κάτω των 3,5 τόνων. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξανακεντραριστούμε, να επανέλθουμε στο άξονα του πολιτικού μας έργου και στο επίκεντρο των εργασιών της Επιτροπής μας, γιατί έχουμε αποκλίνει κάποιους. Στα πλαίσια της διενέργειας του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σέρκα, αλλά για μισό λεπτό παρακαλώ κύριε Σέρκας. Ε, μάλιστα. Δεν θέλω να υπερασπίσω μια θέση. Απλώς να διευκρινίσω το κείμενο της οδηγίας. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι μάλλον δεν διάβασαν προσεκτικά την οδηγία. Γιατί έγινε λόγος για το χρόνο που αφιερώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι σε διοικητικέ διατυπώσει. Αυτό ο χρόνο εργασία είναι εκτό τη οδηγία. Όταν είπαμε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται στο σπίτι του, αν, ε, αν ασχολούνται με το Ιντερνετ, η οδηγία αφορά μόνο τη χειρονακτική εργασία εκφόρτωση των φορτηγών και δεν εμπίπτουν οι διοικητικέ διατυπώσει. Τώρα ξαναρχίστε τη συζήτηση. Ξαναζήτησε το λόγο και η κυρία Χάρκιν. Μα είναι γεγονό, λέει ο κύριο Σέρκα. Ναι, αλλά ο καθένα ερμηνεύει διαφορετικά τα γεγονότα από ό,τι φαίνεται. Τώρα ξαναζήτησε το λόγο η κυρία Χάρκιν, ξαναζήτησε το λόγο ο κύριο Ορή. Ε, πού θα σταματήσουμε. Θα ξαναρχίσουμε με τι ερμηνείε προσωπικέ του καθενό για τα γεγονότα. Θα σα πω λοιπόν και αναλαμβάνω εδώ το λόγο μόνη μου για να σας πω πως ερμηνεύω εγώ τα γεγονότα. Ο κύριος Σόρι. Δεν θέλω να πάρω το λόγο. Πρόκειται για διαδικαστικό θέμα. Βλέπω ότι μας μένει λίγος χρόνος και ενδεχομένω θα έπρεπε να ακούσουμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, προτείνω να ακούσω την άποψή τους. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συμβουλή Ήθελα απλώς να θέσω και μία ερώτηση ακόμα στην κυρία Μπάουερ και μετά να ζητήσω από την Επιτροπή να πάρει το λόγο ε, και μάλιστα θα τους έκανα και, θα έκανα και μία ερώτηση συγκεκριμένη στην Επιτροπή, που δεν έκανε κανένας συζητητής, κανένας ε, ε, βουλευτής. Λοιπόν, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε στην έκθεση αυτή το πνεύμα και το γράμμα της ε, νομικής γνωμοδότησης της 30 Δεκεμβρίου 2009 όταν εμείς ζητήσαμε τη γνώμη της νομικής μας ε, υπηρεσίας ε, σχετικά με τη θέση ισχύ του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002-15. ξεκινώντας από την 23η Μαρτίου. πρέπει να πω ότι δεν συμμερίζομαι όλα τα σχόλια τα οποία ε, ακούστηκαν. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως, ε, εάν όλοι ασχολούνται με την κυρία Μπάουερ και με τη δυσκολία που αντιμετωπίζει, θα μπορούσαν να πούν απλώς συμφωνούμε με την ε, εκδοχή της κυρίας Μπάουερ και τελειώνει το θέμα. Ακούσαμε επανειλημμένα εκπροσώπους των εργαζομένων του ε, κλάδου και ε, είναι γεγονός ότι ο παλιός εισηγητής άφησε πολλά παραθυράκια ε, έτσι ώστε να ικανοποιήσει κατά κάποιο τρόπο τα αιτήματα των εργαζομένων και γι' αυτό ακριβώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση, εν πάση περιπτώσει. Στρέφαμε προς την Κομισιόν. Πρέπει να πω ότι χτες είχαμε μια, μια διαβούλευση όσον αφορά τις νομοθετικές διεργασίες με την Κομισιόν και το Συμβούλιο, την Ισπανική Προεδρία δηλαδή. Γνωρίζομαι ότι ακόμα δεν ε, έχουμε την, ε, τον αρμόδιο επίτροπο ε, στη θέση του, αλλά από ό,τι φαίνεται το πνεύμα του Επιτρόπου κ. Ταγιάννη θα ακολουθήσει και τον διάδοχό του αλλά παρόλα αυτά ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε και την Κομισιόν να μας πούν λοιπόν οι εκπρόσωποι, να μας πει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν εάν έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον διάδοχο του κ. Ταγιάννη, πώς τον έχει ενημερώσει, ποια είναι η πρώτη άποψη. Αν μπορεί να μας πει δύο πράγματα θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Και πολύ σωστά είπε ο κύριος Ορίου ότι θα πρέπει να επέμβει και η Κομισιόν. Δεν ξέρω εάν εσείς θέλετε, κυρία εισηγήτρια, να απευθύνετε κάποιο ερώτημα στην Κομισιόν πριν σας δώσω το λόγο. Μετά, οπωσδήποτε, εσείς θα έχετε τελευταία το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Αλλά μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι πολύ συγκεκριμένο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Πολύ ωραία. Επομένως, θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Πασκουαρέλη ε, για, από τη Γενική Διεύθυνση Τρένου και μετά η κυρία Μπάουερ θα απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σημείωσα το ερώτημά σας και νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω, αλλά ειλικρινά ενοχλούμε με την έννοια ότι δεν μπορώ να σας δώσω τέτοια απάντηση τη στιγμή που ακόμα δεν έχει καν εγκατασταθεί ο νέος Επίτροπος. Ξέρετε ποια είναι η πολιτική του ομάδα, από, ποια από ποιο πολιτικό σχηματισμό προέρχεται. Νομίζω ότι ήδη είπε κάποια πράγματα στη διάρκεια της ακρόασης ε, στην Επιτροπή σας. Τα γνωρίζετε αυτά. Και έστω και αν ε, δεν αντιμετώπισε ευθέως το ζήτημα αυτό, νομίζω λέγω πως όλοι μπορούν να καταλάβουν προς ε, τον προσανατολισμό του, προς τα που οδηγείται η σκέψη του. Αλλά μη με πιέσετε γιατί θεσμικά ε, πραγματικά δεν μπορώ να σας μεταφέρω την άποψη ενός επιτρόπου ο οποίος ακόμα δεν έχει αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του. Εγώ δεν σας λέω ποια είναι η μελλοντική άποψη του μελλοντικού επιτρόπου. Εγώ λέω εσείς πώς προτίθεστε να ενημερώσετε το μελλοντικό επίτροπο. Αυτό θα κάνω. Και θα συνεχίσω στα αγγλικά. Καταλαβαίνω ότι εδώ φύγονται ορισμένα σημαντικά θέματα αρχής. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής σε ένα πρακτικό πρόβλημα ότι οι κανόνες που έχουμε σήμερα δεν έχουν ερμηνευθεί σωστά και εφαρμοστεί σωστά από τα κράτη-μέλη. Και αυτό έχει δώσει αφορμή στο λεγόμενο φαινόμενο του ψεύδο αυτοαπασχολούμενου. Για ορισμένου ιδιώτε δεν είναι επιλογή αυτό, αλλά αναγκάστηκαν να το κάνουν. Είναι μία κοινωνικά δυσμενής κατάσταση την οποία θα πρέπει να διορθώσουμε για να αποφύγουμε την εκμετάλλευση ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν τις αδυναμίες, τα παραθυράκια, τα ελαττώματα τα οποία δημιουργούνται από την λανθασμένη ερμηνεία των σημερινών κανονισμών. Θέλω να τονίσω ορισμένα σημεία τα οποία έχουν οδηγήσει σε σύγχυση την Επιτροπή η βασική δραστηριότητα των οδηγών, είτε είναι υπάλληλοι είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, είναι το οδήγημα, η οδήγηση. Και ο χρόνος οδήγησης και περιόδων αναπαύσεων ρυθμίζονται από ξεχωριστή νομοθεσία, από έναν κανονισμό ο οποίος ορίζει το ελάχιστο 44 ώρες οδήγησης την εβδομάδα. Και για αυτοαποσχολούμενους και για υπαλλήλους οδηγούς και αυτές οι 45 ώρες καταγράφονται από τον, τα, από το ταχύμετρο, ταχογράφο και ελέγχονται από τους αρμόδιους ελεγκτές, την αστυνομία, την τροχέα, ανάλογα ποια είναι η αρμόδια αρχή. Αυτός ο έλεγχος λειτουργεί σχετικά ικανοποιητικά σήμερα και έχουμε εκθέσεις που μας ε, μεταδίδουν αυτό το μήνυμα. Η οδηγία με την οποία σας σήμερα είναι η οργάνωση του χρόνου εργασίας των οδηγών και συμπληρώνει τους βασικούς κανόνες του χρόνου οδήγησης και θέτει ως μίνιμουμ 48 ώρες. Μιλάμε λοιπόν κανονισμούς που καλύπτουν τρεις επιπλέον ώρες οδήγησης. Τρεις επιπλέον ώρες που καλύπτουν φόρτωση-εκφόρτωση, συντήρηση του οχήματος, δυνατότητα συμπλήρωσης των απαραίτητων εγγράφων, ναι, ναι, ναι, ναι, γενικές διοικητικές ε, γραφειοκρατικές αν θέλετε εργασίες οι οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία Γι' αυτό θέλουμε τρεις περισσότερες ώρες. Όλοι μας είπαν, ε, μας είπαν ορισμένα μέλη ότι αυτά γίνονται στο σπίτι, η συμπλήρωση των εγγράφων δηλαδή, αυτές οι διοικητικές εργασίες, την κουζίνα του οδηγού. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Αυτές οι τρεις επιπλέον ώρες καταχωρούνται στο ταχογράφο. Και ο ταχογράφος αυτός δραστηριοποιείται αυτόματα, ξεκινάει να λειτουργεί και να καταγράφει αυτόματα όταν κινηθεί το φορτηγό. Όχι όταν είναι στάσιμο και ο οδηγός έχει βγει έξω και ζητεί από κάποιον να υπογράψει τα έγγραφά του. Ούτε όταν συντηρεί, ελέγχει τα λάστιχα ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχουν επίσης και άλλα συστήματα που πρέπει να πιέσει ε, τον ταχογράφο, να πιέσει ένα κουμπί για να λειτουργήσει ο ταχογράφος. Ο υπάλληλο λοιπόν έχει μεγάλο συμφέρον να πιέσει το κουμπί, διότι δεν θέλει να δουλέψει παραπάνω ώρες. Πρέπει να δείξει τον εργοδότη του πόσε ώρε έχει δουλέψει. Ο ιδιώτη, ο αυτοαπασχολούμενο, δεν έχει αυτό το συμφέρον. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό πρόβλημα. Πώς θα εφαρμοστεί η οδηγία χρόνου εργασίας στους αυτοαπασχολούμενους. Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ελέγχου των ωρών εργασίας ή οδήγησης, αν θέλετε, των αυτοαπασχολούμενων. Γι' αυτό ο, ο σωστός, ο πραγματικός αυτοαπασχολούμενος πρέπει, πιστεύω, να έχει την ελευθερία να οργανώσει τη δουλειά του όπως είναι καλύτερη για αυτόν. Η Γενική Οδηγία αναφέρει πολλά για τους ιδιώτες αυτοαποσχολούμενους. Τώρα, εάν ορίσουμε τους ψεύδο αυτοαπασχολούμενους ότι είναι πραγματικά οι υπάλληλοι εργαζόμενοι που θα πρέπει να εμπίπτουν στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, τότε θα έχουμε λύσει και το, το πραγματικό πρόβλημα που κρύβεται πίσω από αυτούς τους ορισμούς εισαγωγικά. Η τροπολογία λοιπόν που έχει υποβληθεί έχει ως στόχο τον πιο αυστηρό ορισμό των αυτοαπασχολούμενων και αν εφαρμοστεί σωστά και πάλι επιμένω ότι αυτό εξαρτάται από τον τρόπο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας. Το βασικό πρακτικό πρόβλημα ε, της οδηγίας αυτής ε, θα έχει λυθεί. Το πρακτικό πρόβλημα. Λέω λοιπόν στα μέλη αυτά τα οποία ανέφεραν το θέμα της οδικής ασφάλειας. Και εγώ είμαι υπεύθυνο για την οδική ασφάλεια στην Κομισιόν. Προετοιμάζοντα λοιπόν αυτή την νομοθετική ρύθμιση, έχουμε επισταμμένω εξετάσει το θέμα αυτό, έχουμε διαβουλευθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους, τους αρμόδιους, ε, κοινωνικούς εταίρους κλπ. Και δεν έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε οριστική απόφαση για το ποσοστό ευθύνης που έχουν η αυτοαπασχολούμενοι στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Δεν έχουμε καταφέρει να ορίσουμε ποιο ποσοστό οδικής ασφάλειας, συμβολής της οδικής ασφάλειας, αναλογεί στους αυτοαπασχολούμενους. Είναι γεγονός ότι τα στατιστικά στοιχεία, είτε θέλετε ατυχημάτων είτε ασφάλειας, δεν κάνουν ένα ειδικό διαχωρισμό του ποιος φέρει το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης. Αν είναι δηλαδή αυτό ή υπάλληλο. Οι κανόνες αυτοί ε, αναφέρονται και στους, ε, στα φορτηγά τα οποία έχουν ε, βάρος λιγότερο από 3,5 τόνους. Οι οδηγοί αυτών των μικρότερων φορτηγών, κάτω των 3,5 τόνων, υπόκεινται ήδη στη διατάξεις της Γενικής Οδηγίας Χρόνου Εργασίας, διότι δεν καλύπτονται από την ή, τις, τους, ειδικούς, τους, γενικούς κανονισμούς, τους κανονισμούς αλλά καλύπτονται από τη Γενική Οδηγία Χρόνου Εργασίας. Και δει μόνο οι υπάλληλοι. Μόνο οι υπάλληλοι υπόκεινται στη Γενική Οδηγία αυτή. Οι υπάλληλοι οι οποίοι οδηγούν φορτηγά κάτω από 3,5 τόνους. Και όχι αυτό, οδηγοί που οδηγούν, ε, ε, που κάνουν μεταφορές πιτσών σε μικρά φορτηγά. Κάνουμε μία μελέτη λοιπόν και αν ε, τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείξουν ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι, τότε θα το εξετάσουμε. Ε, δεν μπορούμε όμως ε, να κάνουμε ξαφνικά την εισαγωγή του ορισμού του οδηγού φορτηγού μικρού για πίτσες σε ένα τμήμα της νομοθεσίας, δηλαδή να κάνουμε μια ειδική αναφορά μόνο σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε την κυρία Μπάουρ και υποστηρίζουμε την έκθεσή της, την ευχαριστούμε πολύ και χωρίς να δεν είναι δυνατόν ε, χωρίς μεγάλη προσπάθεια να επιτύχουμε ένα συμβιβασμό. Εάν μπορούμε να ελέγξουμε αυτούς τους τρεις τρεις περισσότερες ώρες που ζητάμε των αυτοαπασχολούμενων που με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργήσει υπερβολικό διοικητικό φόρτο, τότε είμαστε πρόθυμοι να το συζητήσουμε. Μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε όμως να βρούμε τρόπο να, βολέψουμε αυτές τις τρεις παραπάνω ώρες ε, χωρίς μεγάλο ε, διοικητικό κόστο. Αν μπορέσουμε τότε εντάξει είμαστε σύμφωνοι να το καταφέρουμε. Εφόσον όμως δεν έχουμε βρει λύση δεν θέλουμε να το θίξουμε, δεν θέλουμε να το πειράξουμε και πιστεύουμε ότι η πρόταση την οποία έχουμε υποβάλει είναι η πρώτη πρακτική. Η πιο πρακτική, η πιο σωστή. Τώρα για τις τροπολογίες της κυρία Μπάουερ, στην τροπολογία 9 αναφέρεται στη συμβολή των κοινωνικών εταίρων για την εφαρμογή και την, για την υλοποίηση και τη συμμόρφωση. Αυτό ήδη υπάρχει. Στην παρούσια οδηγία, άρθρο 13, ε, αναφέρεται υποβολή, υποχρέωση υποβολής εξέσεων στην Κομισιόν μετά από την διαβούλευση και των δύο πλευρών των, της, ε, του τομέα. Και εκτός από αυτό έχουμε μία μικρή συντακτική αλλαγή που, που θέλουμε να γίνει. Σας ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στην συζήτηση αυτή στις επόμενες συνεδριάσεις. Κυρία Μπάουερ, δεν νομίζω ότι μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και τα σχόλια, αλλά φαντάζομαι κάτι θα έχετε να πείτε, γι' αυτό σας δίνω το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή συζήτηση τη της εκθέσεώς σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα αρχίσω από την παρατήρηση της κυρίας Χάρκιν που είπε να ρίξουμε μια ματιά στις μελέτες επιπτώσεων που εκπονήθηκαν προκειμένου να προταθεί η αναθεώρηση της οδηγίας. Οι μελέτες επιπτώσεων διευκρινίζουν ότι η κόπωση εξαρτάται όχι μόνο από το ωράριο εργασία, αλλά και από την ποιότητα του ύπνου, από την ε, ημερήσια περίοδο, από την οικογενειακή κατάσταση του οδηγού μεταξύ άλλων και είμαι πεπισμένος ότι ένας ε, οδηγός που βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου είναι κουρασμένος ήδη από το πρωί ε, όπως και ένας οδηγός που έκανε για τρεις ώρες ε, φόρτωση-εκφόρτωση εμπορευμάτων. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα και να ελέγχουμε και τις ε, ώρες ε, ανάπαυλας για να δούμε πώς τις πέρασε ο οδηγός και να δούμε τι έκαναν στο διάλειμμα τους ή τι κάνουν στο χρόνο αναψυχής τους, αν έκοβαν ξύλα ή αν έβλεπαν τηλεόραση. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και στατιστικά στοιχεία που υποστηρίζουν τη θέση της. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία λένε ότι ο κάματος, η κόπωση ε, είναι υπεύθυνη για το 0,6% των ε, τροχαίων ατυχημάτων. Δεν υπάρχει βέβαια διάκριση ανάλογα σε αυτό που ή μη. Ζητούμε αναλογικότητα στην εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Και σας διαβεβαιώ ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλω να παρακάμψω το θέμα της οδικής ασφάλειας. Απλώς είπα ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, προκειμένου να καλύπτει και τους αυτοαπασχολούμενους, κατά τη γνώμη μου ήταν ακατάλληλη λύση και για το 2002 και για σήμερα. Από το 2002 και μετά είχαμε θεαματικές εξελίξεις. Είχαμε πολύ περισσότερη ρύθμιση οδηγίες ε, που ρυθμίζουν ε, το έργο του οδηγού. Είχαμε την 561 του 2006 οδηγία για παράδειγμα, αλλά και άλλες. Οπότε άλλη κατάσταση έχουμε σήμερα από αυτή που είχαμε το 2002. Και νομίζω ότι καταρχήν η απόφαση του 2002 δεν ήταν σωστή. Μετά από τη συζήτηση αυτή, δημιούργησε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση του κοινωνικού ντάμπινγκ με το χρόνο που αυτό αποσχολούμενος αφιερώνει στη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτηγού του. Η οδηγία ασχολείται μόνο με το θέμα των οδηγών, ενώ το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο. Οπότε δεν υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού μεταξύ των δύο. Σέβομαι τον κύριο Σέρκας και εκτιμώ ιδιαίτερα την προσήλωσή του στα θέματα της ρύθμισης του ωραρίου εργασίας, αλλά δεν νομίζω ότι το ΔΕΚ εξέδωσε νομολογία τέτοια όπως μας περιγράψατε. Σήμερα η κατάσταση ε, διαφέρει για τους μισθωτούς και για τους αυτοαπασχολούμενους. Κύριε Ρες, και εγώ είδα τη γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας. Εκεί αναφέρεται η παρούσα κατάσταση και διευκρινίζεται ότι υπάρχουν διατάξεις που ισχύουν και για τους αυτοαπασχολούμενους. Και αυτό θέλουμε να αλλάξουμε σήμερα. Τώρα, για να προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Τόμας Μαν. θέλω να πω. Είπατε κύριε Μαν καταρχήν ότι δεν είναι σκόπιμο να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή των ψηφιακών ταχογράφων στους υπαλλήλους που κάνουν παραδόση φαγητού κατοίκων, πίτσας και άλλων. Δεν νομίζω ότι εμείς οι Επίτροπός μας ε, ε, είμαστε αρμόδιοι να ρυθμίσουμε αυτά τα όρια. Συζήτησα το ζήτημα αυτό και με τον κύριο Χιούς και το συζητήσαμε και με τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών και αποφασίσαμε να ορίσουμε το όριο στο 2,8 τόνους. Αλλά αυτή είναι αδύνατο στην οδηγία αυτή, γιατί όλες οι ευρωπαϊκές ε, διατάξεις προβλέπουν ε, τους 3,5 τόνους ως όριο. Αλλά και όλες οι διεθνείς συμφωνίες έχουν αυτό το όριο των 3,5 τόνων. Οπότε χαιρετίζω την πρόταση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα εκπονήσουν μια μελέτη για το θέμα αυτό. Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Να γίνει μια μελέτη για να αξιολογηθεί η κατάσταση και μάλιστα τις προάλλες που συζητήσαμε αυτό το θέμα, πολλοί επισήμαναν την ανάγκη περαιτέρω μείωση αυτού του ορίου βάρους για τα φορτηγά. Αλλά αυτό δεν γίνεται στην παρούσα οδηγία. Πολλοί συνάδελφοι επιβεβαίωσαν ότι οι οδικές μεταφορές πολύ συχνά πραγματοποιούνται από μικρά οχήματα, κάτω των 3,5 τόνων. Ίσως η Επιτροπή Μεταφορών θα έπρεπε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης, θα ήθελα να πω ότι όλες οι επιχειρήσεις, είτε είναι μικρές, είτε μεσαίες, είτε μεγάλες, θα καλύπτονται από την διάταξη αυτή. Κατά τη γνώμη μου, παραλαμβάνω, το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία δεν θα πρέπει να επεκταθεί και στου αυτοαπασχολούμενου. Κύριε Χέντελ, είπατε ότι είναι αδύνατον να ελέγξουμε τι γίνεται στο δρόμο συνέχεια. Οι επιθεωρητές εργασίας είναι αυτοί που θα ελέγξουν το θέμα αυτό και στις, στους ελέγχους που γίνονται στο δρόμο, το, το μόνο που μπορούμε να επαληθεύσουμε είναι το, το νούμερο που περιλαμβάνει ο ψηφιακός ταχογράφος. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρίνησε τι είναι εφικτό και τι όχι ως προς τον έλεγχο. Αυτά κυρία Πρόεδρε, αυτές ήταν οι απαντήσεις μου και περιμένω τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπάουερ. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 5 ε, Φεβρουαρίου στις 2 το απόγευμα στις 12 το μεσημέρι, συγγνώμη, και επίσης 4 Μαρτίου η Επιτροπή Μεταφορών θα μας δώσει ε, θα μας έχει δώσει ήδη τη γνωμοδότησή της και επομένως θα ψηφίσουμε στις 16 και 17 Μαρτίου. Επόμενη συνεδρίαση στις 22 ε, Φεβρουαρίου υπό την Προεδρία της κυρίας Λίν. Δεν ξέρω εάν τώρα θα πρέπει να πατήσετε αυτό το ειδικό κουμπάκι στον ταχογράφο σας και αν θα είναι ώρα εργασίας, αλλά πάντα